Eh, λοιπόν, η Βαρόνια Άστον συνάδελφοι, η ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακριβή στην ώρα τη. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια κυρία τόσο αξιότιμη να περιμένει. Την καλωσορίζουμε εκ μέρου όλων σε αυτή τη συνάντησή μα. Ε, είναι η δεύτερη φορά στην οποία πρωταγωνιστεί στο διάλογο μεταξύ μας. Αν και με τη Βαρόνια Άστον υπήρξαν και άλλες περιστάσεις όπου συναντηθήκαμε κάπως πιο άτυπα, αλλά ήταν εξίσου καρποφόρες οι συναντήσεις. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η συνθήκη της Λισαβόνας, ε, το ξέρει και καλύτερα από όλους η κυρία Διάστον, ανέθεσε ευθύνε στη θέση της. Και για ανεπομιστή τις ευθύνες δεν χρειάζεται μόνο να καινοτοποιήσουμε τη μέθοδο εργασίας, αλλά να τις διαθέσουμε και μέσα επιμελητίας και πόρους για να μπορέσει να εκτελέσει το καθήκον της. Μπορώ να πω εν ονόματι όλων των συναδέλφων ότι αυτό το Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα η δική μας Επιτροπή την υποστήριξε στην προσπάθεια να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης η οποία να μπορεί να πλαισιώνει τις πολιτικές της δράσης στο διεθνές προσκήνιο. Χρειάζονται μέσα κατάλληλα για τις φιλοδεξίες που έχουμε θέσει σε αυτό το πλαίσιο και τις προοπτικές που ε, δημιουργούνται και προσδοκίες που έχουμε όλοι. Τώρα είμαστε στη φάση στην οποία θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο των σχέσεών μας Πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένας πολιτικός καρποφόρος διάλογος όσον αφορά το ρόλο της ενώσεως, ποιες είναι οι προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης στο διεθνές προσκήνιο, ποιες είναι οι προτεραιότητες που πρέπει να κατευθύνουν τις δράσεις μας και βεβαίως ποια είναι τα αναγκαία μέσα για να επιδιωχθούν αυτοί οι σκοποί. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο όπως συμφωνήσαμε, κυρία Άστον, σήμερα να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε το διάλογό μας στο μέτρο του δυνατού επί των προτεραιοτήτων που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ακροθυγώς, αλλά δεν θα ήθελα να αναφέρουμε πολλά σημεία για να εμβαθύνουμε στα διάφορα σημαντικά θέματα, όπως είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, ε, ποια θα μπορούσε να είναι η πολιτική της Ενώσεως ε, όσον αφορά το ευαίσθητο θέμα των σχέσεων με το Ιράν, η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι ήταν ένα από τα βασικά σημαντικά σημεία της συζητήσεως που έλαβε χώρα εχθές στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ενώσεως. Θα το επαναλάβουμε και εδώ. Τα προβλήματα τα σχετικά με τη δράση της Ενώσεως στο κέρας της Αφρικής και οι σχέσεις με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Αυτό το τελευταίο είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα προσφυλές σε εσά και σε εμάς φυσικά. Δεν χρειάζονται νομίζω άλλες εισαγωγές για να ξεκινήσουμε τη συνάντηση μαζί σας. Βαρώνει, έχετε το λόγο και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ μαζί μας, να είσαστε μαζί μας και σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι πολύ ικανοποιημένη που είμαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έλεγα πάντα ότι είναι σημαντικό να γίνεται τακτική ε, ανταλλαγή απόψεων και είναι μια δυνατότητα για μένα να ακούω τις ανησυχίες των ε, βουλευτών και ιδιαίτερα να ακούσω τα μέλη αυτής της Επιτροπής και μια ευκαιρία για μένα ίσως να διερευνήσω περαιτέρω κάποιο από το έργο που, στοιχεία του έργου που τελούμε. Θα είμαι σύντομη όσον αφορά τις παρατηρήσεις μου διότι ενδιαφέρομαι στο, να ακούσω το διάλογό μας, να συμμετάσχω στο διάλογό μας, αλλά θα ήθελα να αναφέρω κάποιους συγκεκριμένους τομείς ε, που εσείς Πρόεδρε θίξατε, σημεία που θα ενδιαφέραν τους περισσότερους και θα ήθελα να τα αναφέρω σήμερα. Όταν ξεκίνησα είπα ότι θα έχω τρεις βασικές προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα είναι η υπηρεσία εξωτερικής δράσεως, η σύστασή της, και χάρη στο Κοινοβούλιο, ευχαριστώ πολύ του Ευρωβουλευτέ για την υποστήριξη και τη βοήθεια και τον προσανατολισμό, φτάσαμε στο σημείο, λέγω, όπου θα μπορέσουμε να μπούμε στην επιχειρησιακή φάση. Θα λειτουργήσει η υπηρεσία. Δεύτερη προτεραιότητα είπα ότι θα είναι η γειτονία, η πολιτική γειτονία και υποψιάζομαι ότι κάνα δύο συνάδελφοι θα ήθελαν να το εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Ήθελα για λίγο να εστιαστώ επ' αυτού, διότι προφανώς ε, ταξίδεψα, πήγα στην Ουκρανία βεβαίως, στη Ρωσία, στη Γεωργία, στα Δυτικά Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο και θα έχουμε τη Διπουργική Σύνοδο της Ανατολικής Γειτονία σύντομα. Αν ήθελα να υπογραμμίσω μια πτυχή τη πολιτικής μας της γειτονία, θα ήταν η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο η απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων να στείλει τη σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι κάτι σημαντικό για τη Σερβία. Ε, θέλουμε να γίνουν κινήσεις και για το κοσυφοπεδίο ε, να γίνει και εκεί αποτίμηση των πρόοδων που έχουν επιτευχθεί. Ξέρω κάποιοι βουλευτές πέρασαν μεγάλο χρονικό διάστημα στα Δυτικά Βαλκάνια και Κωσυφοπέδιο και Σερβία, ιδιαίτερα πρόσφατα. Λοιπόν, η άλλη προτεραιότητα, όπω είπα, είναι η στρατηγική εταίρη και για μένα αυτό είναι ουσιαστικό, σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει από μόνη τη να καθορίσει ε, τι μορφή θα ήθελε να έχουν στο μέλλον αυτέ οι σχέσει. Ε, πέρασα πολύ χρόνο, δικό μου χρόνο, συζητώντα το θέμα με του εταίρου μα, προφανώ με τη Χίλαρη Κλίντον στι Ηνωμένε Πολιτείε. Με τον, ε, πήγα στην Κίνα και είδα τον κύριο Νταγκβό τον Αύγουστο για τον Πρωθυπουργό Γιάνγκ και είδα και τον κύριο Λαύροφ ε, στην Ρωσία, συναντούμε τακτικά και είδα και τον Πρωθυπουργό Κρίσνα στην Ινδία και εκεί εξετάσαμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα το στρατιωτικό και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε συνεργασία με την Ινδία. Λοιπόν, βασικά στοιχεία για τους εταίρους μας στρατηγικούς. Θα έλεγα ότι οι εταίροι μας έχουν μια σαφή εικόνα σχετικά με το τι θέλουν να υπάρξει στη σχέση αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ο κόσμος έτσι όπως έχει δημορφωθεί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχουμε, μας δημιουργεί με δυνατότητα να είμαστε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά το τι θέλουμε να πετύχουμε από τις εταιρικέ σχέσεις που έχουμε. Και τι ξεκινήσαμε. Ε, καλέσαμε επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων να μου δώσουν εντολή να επεξεργαστώ ιδέες για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις με τους στρατηγικούς εταίρους να δούμε τι σχέση θέλουμε να έχουμε μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Ε, θα αναφερθώ στο, γενικό, στο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου ε, ποια θα είναι αυτά τα σχέδια. Τα μέλη της Επιτροπής σας θα ήθελαν να εστιαστούν ενδεχομένως σε διαφορετικούς στατηγικούς εταίρους, ίσως σε διάφορες πτυχές του σχετικά, σχετικά με τις σχέσεις μας με αυτούς τους εταίρους μας στο μέλλον. Βεβαίω, ε, εστιάζονται οι προσπάθειε και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Τον Ιούλιο πήγα στην Καμπούλ και πήγα στη διάσκεψη που έλαβε χώρα εκεί που δημιούργησε τα νέα προγράμματα εθνικών προτεραιοτήτων. Όταν συναντήκαμε τον πρόεδρο Καρζάη, του ξεκαθάρισα ότι καταρχά η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι υπάρχει μακροχρόνιο έργο που πρέπει να επιτελεστεί και δεύτερον θα ήταν σημαντικό ε, να συμμετάσχει όλη η κοινωνία, κυρίως οι γυναίκες σε αυτή την προσπάθεια. Το πρωί της διασκέψεως συναντήθηκα με τη Χίλαρη Κλίντον και κάποιες Αυγανές γυναίκες. Εκεί συζητήσαμε ένα ολόκληρο φάσμα θεμάτων που τους ενδιαφέρε μικροχρηματοδότηση, οικονομική ανάπτυξη, παιδεία και υποψηφιότητα σε εκλογές. Αυτό είχε λάβει χώρα πριν από τις ε, εκλογές. Αυτές οι γυναίκες, κατά την άποψή μου, ε, ήταν κρισίμου σημασία για τη μελλοντική κατεύθυνση του Αφγανιστάν και είναι πολύ σημαντικό να στέλνουμε αυτό το μήνυμα ότι θα πρέπει οι γυναίκε να συμμετέχουν συνεχώ στι διάφορε διαδικασίε που θα λαμβάνουν χώρα εκεί. Και ξέρω ότι διάφοροι εδώ γνωρίζουν πολλά για το Αφγανιστάν και σίγουρα θα επιστρέψουμε στο μέλλον στο ζήτημα αυτό. Όσον αφορά το Πακιστάν, ε, πρόσφατο γεγονότο ήταν οι φίλοι του Δημοκρατικού Πακιστάν, προείδευσα εκεί με τον Υπουργό Καράση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς πώς βλέπουν τους 17 τομείς και προσπαθούν να καθορίσουν την καλύτερη χρήση των πόρων της διεθνούς κοινότητας και τους δικούς τους πόρους, ώστε να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα αποτελέσματα των πλημμυρών, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη που θέλουν να πετύχουν. Και βέβαια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το εμπόριο, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Πακιστάν. Και πρέπει να σας πω ότι η αντίδραση του Πακιστάν, και θα ήθελα να στείλω αυτό το μήνυμα προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Πακιστάν έλεγα αναγνώρισε τη σημασία όλων αυτών και ήθελε να θεωρηθεί αυτό ότι είναι σημαντική κίνηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που τους υποστήριξε. Όχι μόνο αμέσως τώρα αλλά και στο μέλλον. Λοιπόν, θα στραφώ τώρα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που όλοι περιμένουμε με ανησυχία να δούμε ποια πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί τώρα. Ε, έχω τακτικές επαφές με τον κ. Μίτσελ και Είδα ότι είναι πάρα πολύ δραστήριο σε αυτό το τομέα, συνεργάζεται και με του Ισραηλινού και του Παλαιστινίου, προσπαθώντα να βρει μια διέξοδο από το τέλμα που βρίσκονται τώρα. Είμαι στην περιοχή εδώ και τις τέσσερι εβδομάδε και είχα κατηδίαν συναντήσει με τον πρόεδρο Αμπά, τον πρωθυπουργό Φαγέτ και τον πρωθυπουργό Νετανιάχου ήθελα να πω και τον γερουσιαστή Μίτσελ τον ίδιο. Ε, είναι σαφέ ότι η πραγματική επιθυμία υπάρχει για πρόοδο, αν μπορούμε να βρούμε μια διέξοδο ε, σε όλα τα θέματα που έχουμε, το θέμα του ε, μορατόριου. Εγώ του είπα ποια είναι η θέση μα. Επανειλημμένα σε κάθε τηλεφώνημα, σε κάθε επίσκεψη έλεγα ποια είναι η θέση μα. Και χτε συζητούσα το θέμα με τον Ιορδανό Υπουργό Εξωτερικών. Διαδραματίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο. Υποστηρίζουμε τι προσπάθειε και εξασφαλίζουμε το ότι το κουαρτέτο είναι ενεργό ε, προωθούμε την ε, προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ενώσης, επί της οποίας συμφωνούμε για υποστήριξη του μέλλοντος, για υποστήριξη της ανάπτυξης του Παλαιστινιακού κράτους και θέλουμε εκείνοι να μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως στις διαδικασίες για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο μέλλον. Πρέπει όμως ε, να κάνουμε περισσότερο για να, όταν προχωρήσουν συνομιλίες για να υπάρξει και συμμετοχή της διεθνούς κοινότητας. Όταν σκέφτομαι βέβαια τη Μέση Ανατολή, σκέφτομαι αναπόφευκτα και το Λίβανο και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συζητήθηκε το θέμα όταν συζητήθηκε η υποστήριξη τη σταθερότητα τη κυβερνήσεω εκεί και τονίστηκε η σημασία των όσων είπε ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ όσον αφορά το ειδικό δικαστήριο. Οι συνάδελφοι ενδιαφέρονται επίση και για το Ιράν και θα γνωρίζετε βεβαίω ότι επίσημα έστειλε επιστολή στον Δ. Τζαλίλη που είναι ομόλογό μου να προτείνω να ξεκινήσουμε ε, στην Βιέννη τον Νοέμβριο. Ε, περιμένω την απάντησή του, αλλά πάντα ε, έλεγα ότι είναι διτή προσέγγιση. Είναι σημαντικό να πιέζουμε, είναι σημαντικό και να είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του διαλόγου και αυτό το καταστήσαμε σαφές και στη δέσμευσή μας να προωθήσουμε το διάλογο. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Βεβαίω είδαμε το πακέτο που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέτρα, ε, ούτω ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε την πίεση. Και το, με τον Μπάντι συναντήθηκα, ε, πήρε το Νόμπελ Ειρήνη, ε, κάνει προσπάθειε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, εντυπωσιακή και εξακολουθούμε να έχουμε επαφή. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι τι γίνεται έξω από τι ακτέ τη Σομαλίας με την αποστολή Αταλάντη και πέρα από αυτό το ποια είναι η συνολική προσέγγιση στην προσπάθεια που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που οδηγούν σε πειρατεία στις ακτές. Ήμουν στην Αφρική για δεύτερη επίσκεψη στην περιοχή, συμπρόεδρος μιας συνεδριάσεως, εξετάζοντας το πώς η αφρικανική ηγεσία μπορεί να εξασφαλίσει καταρχάς διαμόρφωση στρατηγικής για τη Σομαλία, να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε ε, την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή με τη βοήθεια του ΟΗΕ και θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ οι θαλάσσιες διώδη για να συνεχίζεται η διέλευση του εμπορίου, να μπορούν να παραδίδονται τρόφιμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, να εφαρμόζουν τα προγράμματα παραδόσεως τροφίμων και τα πληγέντα κράτη θα πρέπει να βοηθηθούν να είναι πιο αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της πειρατείας που μαστίζει τις ακτές τους. Νομίζω ότι πήρατε μια γεύση όλων των θεμάτων ε, που θα συζητήσουμε σήμερα. Είμαστε πολύ δραστήριοι και με τη δημιουργία της υπηρεσίας θα μπορέσουμε να παρέχουμε καλύτερες ακόμα υπηρεσίες. Πάνω απ' όλα θέλω να πω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, ε, έχει αντιπροσωπείς επιτόπου και έχει σημασία το έργο που κάνουν εκ μέρους μας όλοι στον κόσμο και γι' αυτό με αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να σε ευχαριστήσω όλους. Σε ευχαριστώ Βαρόνι. Θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ε, με την ευχή να βγουν Ανατολισμή σε μία προς εξέταση προτάσεις και συστάσεις που θα βοηθήσουν το πολύτιμο έργο σας. Θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές. Τρία λεπτά ο καθένας για τους συντονιστές και μετά θα πρέπει να μειώσουμε σε λιγότερο χρόνο για τις απλές παρεμβάσεις. Ο κύριος Σαλανφράγκα, συντονιστής του ΕΛΚ, έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τη Βαρόνια Άστον για την παρουσία της στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω αν όχι με μια ανθοδέσμια όπως το κάναμε στην Ολομέλη. Την ευχαριστούμε παρόλα αυτά για την προσπάθεια που κάνει να έρχεται τακτικά στη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. Και θα ήθελα να τη συγχαρώ, αλλά και να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για την ψηφοφορία στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα υπέρ τη σύσταση υπηρεσία εξωτερική δράση. Και ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβει σάρκα και ωστά θα γίνει μια πραγματικότητα που θα εκπροσωπεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ξεφύγω λίγο από τον κατάλογο των θεμάτων που μα παρουσιάσετε κυρία, κύριε Πρόεδρε, και θα θέσω μια ερώτηση για την Κούβα. Γιατί το Συμβούλιο τη Δευτέρα έλαβε την απόφαση να μην τροποποιήσει τη θέση του, αλλά να ε, ξεκινήσει διερευνητικές ε, διαπραγματεύσεις εν ώψη μιας πιθανής προσέγγισης. Σε σχέση λοιπόν ε, με αυτή την τροπή στο Συμβούλιο, συμμερίζεστε τις διακηρύξεις του προκατόχου του κυρίου Σολάνα ότι δηλαδή η κουβανική κυβέρνηση πρέπει να μην περιοριστεί μόνο στο να απελευθερώνει πολιτικούς κρατουμένους και να τους απελάβει από τη χώρα. Θα πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Επίση, ο Κουβανό ΥΠΕΞ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα δικά τη προβλήματα, στα του οίκου τη, από ότι να σκέφτεται μία προσέγγιση με βάση την παρούσα θέση του Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε τη συνθήκη και την ανάγκη σύγκληση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη λήψη υπόψη των ψηφισμάτων. Φυσικά γνωρίζετε τα τελευταία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της Κούβας, μετά το θάνατο του Ορλάντο Θαπάτα και την απόφαση της συνδιάσκεψης των Προέδρων μετά τις ψηφοφορίες Επιτροπές Εξωτερικών και Ανάπτυξης να δώσουμε το βραβείο Ζαχάρος στον Κιγέρμο Φαρίνιας. Είστε έτοιμοι να επέμβετε κυρία Στον ώστε να μπορέσει ο κύριος Φαρίνιας να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ που του απένιμαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και να ασκήσει το θεμελιώδη του δικαίωμα εξόδου και επανεισόδου στην πατρίδα του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα και μάλιστα διότι σεβαστήκατε και το χρόνο που σας διετέθη. Βίγγενινγκ για τρία λεπτά. Κύριος Βίγγενιν. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας κυρία Άστον. Επιτέλους περνάμε από την διαμόρφωση των δομών και των διαρθρώσεων στην πραγματική χάραξη και ανάπτυξη των πολιτικών. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό. Τώρα, μια στρατηγική ερώτηση για τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Ποια είναι η γνώμη σας ε, για το πού θα πρέπει να στηρίζονται αυτές οι στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Γιατί για πολλούς από εμά, οι χώρες με τις οποίες συζητούμε σίγουρα είναι εταίροι που θα πρέπει να έχουν στρατηγική σημασία και έχουν τις δυνατότητες, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών. Και όταν ακολουθούμε μια συγκεκριμένη πολιτική απέναντί τους, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μετά τη Λισαβόνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει διαφορετικό ρόλο, να γίνει ηγετική δύναμη για πολλά θέματα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ακρίβεια ποιοι είναι οι στόχοι μας απέναντι στους στρατηγικούς αυτούς εταίρους μας. Δηλαδή θα έχουμε μεγαλεπίβολο στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης, για παράδειγμα, ή μήπως ε, προτιμούμε μια ρέγγιση μια βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών, την ε, βελτίωση του επενδυτικού κλίματος Μπορούμε να μιλούμε για κοινέ αξίες ή θα πρέπει απλώς ε, να θεσπίσουμε κάποιους κοινούς στόχους για την υλοποίηση με τους ε, εταίρους μας. Μπορούμε να έχουμε κοινούς στόχους με όλους τους εταίρους, τους ίδιους στόχους. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν και στην Επιτροπή μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ενδιαφέρει η γνώμη σας γιατί είστε είπατε και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Δεύτερο θέμα, είμαι αρμόδιο στην ομάδα μου για το διάλογο Σερβίας-Κωσυφοπεδίου. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το διάλογο που αρχίζει και επαναλαμβάνεται μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Κωσυφοπεδίου και τις εκλογέ. Πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία, προβλέπετε ένα χρονοδιάγραμμα, έχετε κάποια σχέδια πώς θα προχωρήσετε σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό και υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου ε, για την ε, υποβολή υποψηφιότητας ένταξης Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Βίγκενεν. Η κυρία Νέιτς έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Ήπατη Άρμοστη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ε, συνεδρίασή μας και να σας ε, συγχαρώ για τα θέματα που έχετε θέσει μετά από την τελευταία σύνοδο. Να σας συγχαρώ επίσης και να συγχαρώ και τον εαυτό μας που καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνίες και να εγκριθούν όλα βασικά άμα έγγραφα αναφορικά με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, άρα θα μπορέσουν να ξεκινήσει τις εργασίες της υπηρεσία. Έχουμε όμως ε, κάποια ερωτηματικά για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Χτες ε, μιλήσαμε εκτενώς για το θέμα αυτό με τον Επίτροπο Φίλε και ανέφερε μία από τις ανησυχίες σας. Τις παγωμένες σειράξεις, τις παγωμένες συγκρούσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν έχετε κατά νου να, να λάβετε κάποια συγκεκριμένη δράση για να απεγκλωβιστούν, να λυθούν αυτές οι καταστάσεις σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά να τερματίσουμε το στρατιωτικό σκέλος των επιχειρήσεων. Γιατί όλο και πιο σαφές ε, γίνεται ότι δεν πρόκειται να είναι στρατιωτική λύση. Θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα με πολιτικό τρόπο. Δεν ε, έχω φυσικά την προσδοκία ότι θα μας αποκαλύψετε τα πολιτικά μυστικά και τις πολιτικές συνομιλίες που γίνονται για το θέμα αυτό, αλλά ασφαλώς και θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί μέσα Ανατολή φυσικά όλοι θέλουμε να επιτευχθεί μια λύση. Να σας ρωτήσω αν γίνονται επαφές και τι επαφές γίνονται με τους ηγέτες της Λίγκας της Αραβικής, και όλων των χωρών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Και που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξέβρεση ειρηνικής λύσης. Λούνατσεκ για τρία λεπτά, κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ Εξωτερικών, θέλω να σας αποκαλώ. Εγώ μπορώ να χρησιμοποιώ ό,τι λέξεις μου αρέσουν, κύριε Τάνοκ. Έτσι θα σας λέω λοιπόν στο μέλλον. Και εγώ θέλω να σας συγχαρώ που καταφέραμε να περάσουμε τη συμφωνία προκειμένου να ξεκινήσει τις εργασίες της από 1η ε, Δεκεμβρίου η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ωστόσο, όπως ε, ξέρετε, τα θέματα της οικοδόμησης ειρήνης και της διαχείρισης ε, ε, πολιτικών κρίσεων είναι θέματα πολύ σημαντικά και θέλουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να μας πείτε πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε ως ε, εισηγήτρια για το Κωσυφοπέδιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχάς, ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ε, ε θεωρήσεων σε ό,τι αφορά και το Κωσυφοπέδιο. Χτες ε, δόθηκε το πράσινο φως να ξεκινήσει τη διαδικασία στην Σερβία και είναι νομίζω σημαντικό ουσιώδες η Επιτροπή τώρα να δώσει σχετικό χάρτη πορείας και στο κοσυφοπέδιο. Η Αλβανία θα έχει τέτοιες ε, ελευθερίες σύντομα και οι μοναδικοί στην περιοχή που δεν ξέρουν πότε θα έχουν τέτοιες ελευθερίες είναι οι Κωσοβάροι και έχουν κάνει πολλά ξέρετε και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας όλα, σε όλα τα έχουν κάνει. Πριν το καλοκαίρι τους είχαμε πει ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε. Δεν υπάρχει καν στρατηγική ακόμα. Τι θα κάνετε με το θέμα αυτό και το θέμα, το δεύτερο θέμα είναι το θέμα του διαλόγου. Ξέρω ότι υπάρχει ε, θεσμική κρίση στο Κωσυφοπέδιο σήμερα. Αλλά κοιτάξτε, αυτό δεν χρειάζεται να σταθεί εμπόδιο στο διάλογο. Ποιο είναι λοιπόν το χρονοδιάγραμμά σας και πότε θεωρείτε ότι μπορείτε να αρχίσετε να συζητάτε βασικά θέματα. Και τελευταίο ερώτημα για την ε, διαδικασία για την Μέση Ανατολή. Σήμερα το πρωί μου προκάλεσε μεγάλο σοκ ε, οι ειδήσει στη Euronews και αλλού από διαμαρτυρίες ε, Αράβων και Ισραηλινών που διαμαρτύρονταν κατά μιας νέας νομοθεσίας που απαιτεί από οποιονδήποτε θέλει να ε, ονομάζεται Ισραηλινός, να έχει την Ισραηλινή ηθαγένεια, να δηλώνει την πίστη του και στην θρησκεία, το οποίο φυσικά για τους Άραβες Ισραηλινούς είναι ένα θέμα. Ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Βάζουμε ανάμεσα στους συντονιστές αντιπρόεδρο, πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Προβέρα. Για τρία λεπτά. Συγχαρητήρια και ευχαριστώ για την παρουσία σας ε, εδώ, Βαρόνι Άστον. Θα αναφερθώ στην Σομαλία. Από το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δαπάνησε 147 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξει τη στρατιωτική αποστολή τη Αφρικανική Ενώσεω για να σταθεροποιηθεί η χώρα. Αυτό χωρί να μετρήσουμε διάφορε συνεισφορέ που δόθηκαν από μεμονωμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποτελεσματικότητα αυτών των στατευμάτων επιτόπου είναι πολύ μέτρια διότι η πιν ομοσπονδιακή κυβέρνηση μεταβατική κατέχει το προεδρικό ανάκτορο, το αεροδρόμιο το δρόμο μεταξύ των δύο αυτοτόπων περίπου λίγο παραπάνω από 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι στρατός της Αλ-Σαμπάντ και ε, το Ισλαμικό Δικαστήριο εξαπλώνονται σε πολλά μέρη της Σιμαλίας και συνέπεια είναι η αποσταθεροποίηση όλου του κέρατος της Αφρικής. Η μόνη ασφαλής και σταθερή περιοχή εδώ και χρόνια είναι η Σομάλιλαντ που αγνοήθηκε και αμελήθηκε από τη εθνική κοινότητα και κατά θαυματουργό τρόπο βρήκε ισορροπία μεταξύ των διαφόρων φυλών. Τρεις προεδρικές εκλογές έλαβαν χώρα από τον πρόεδρο Εγκάλ μέχρι τον Παρόντα που διεξήχθησαν δημοκρατικά και ειρηνικά. Υπό το φως του γεγονότος ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Αφρικανική Ένωση έχουν ανοιχτή συνεργασία και εταιρική σχέση με την κυβέρνηση της Ομάλιλαντ. τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνω, δεν πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο, αναγκαίο, βαρώνει άστον, να επενδύσουμε πολιτικός και οικονομικός στην Σομάλιλαντ που είναι ένα πρότυπο σταθερότητας για τους άλλους Σομαλούς και μπορεί να είναι ένας διαμεσολαβητής για την κρίση ακολουθώντας τις παραδόσεις των Σομαλών και χωρίς να χρειάζονται αμέτρητες διεθνείς διασκέψεις που είναι δαπανηρές, που γίνονται στη γειτονική Κένια και δεν έχουν αποδώσει μέχρι τώρα και καρπούς ή σημαντικά αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Προβέρα. Το λόγο έχει ο κύριος Τάνοκ για ένα τρίλεπτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θερμό καλωσόρισμα στην Βαρόνια Άστον, τη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να σας συγχαρώ ε, για τα επιτεύγματά σας και για τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσεως, αλλά εγώ θα ζητούσα ε, να υπάρξει ε, δημοσιονομική ουδετερότητα, κάτι που ζήτησα, αλλά υπάρχει λιτότητα σε όλη την Ευρώπη και άρα και σε επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνουμε παράδειγμα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα όσον αφορά την Αφρική που αναφέρθηκαν ακροφυγώ, αλλά ένα δεν αναφέρθηκε. Είναι το Νότιο Σουδάν και το επικείμενο δημοσίφισμα για την ανεξαρτησία θα έρθει εδώ στο εγγύς μέλλον ο Υπουργό Εξωτερικών και ένας από τους Υπουργούς της ε, περιοχής. Υπάρχουν προβλήματα, διορίστηση είχαμε και τη Ρόσλιν Μάρτζ ε, που ε, διορίστηκε από εσά εδώ και μερικές εβδομάδες. Τα πάντα ακολουθούν τον δρόμο του και οτιδήποτε απόφυρα του Προέδρου Μπασίρ να εκτροχιάσει τη διαδικασία θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση τη Ευρωπαϊκή Ενώση και των κρατών μελών τη και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε για να βοηθήσουμε να υπάρξει μια αποστολή παρατηρητών των εκλογών και να τους δώσουμε συμβουλές πώς να διεξάγουν το δημοψήφισμα κλπ. Και, και το άλλο αναφέρεται τώρα στην Αφόρ, Αταλάντα και το κέρας της Αφρικής. Όλοι γνωρίζουμε ότι βασικά η Σομαλία είναι μια χώρα που έχει καταρρεύσει μεταβατική κυβέρνηση, μεταβίας καταφέρει να ελέγξει την πρωτεύουσα. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε, κάνετε περισσότερα για να πάτε σε αυτή την νόση της σταθερότητας, να έχετε σε επαφή με αυτούς στην της σταθερότητας που ε, την τον περασμένο μήνα η Σομάλιλαντ που ήταν ένα βρετανικό προτεκτοράτο κάποτε. Η Σομάλιλαντ διεξήγαγε τις προεδρικές ε, εκλογές, είναι σταθερή, έχει αγνοηθεί, μπορείτε να βρείτε τρόπους χωρίς να αναγνωριστεί, γιατί το 1960 ήταν για μια εβδομάδα κράτος Εγώ πιστεύω αυτό θα ήταν ε, ναι, εκ νέου αναγνώριση πέραν, εκτός από αναγνώριση που έδωσε των ηθική υποστήριξη, διότι βοήθησαν πάρα πολύ σταθεροποίηση, στην προσπάθεια σταθεροποίηση του κέρατος της Αφρικής και τα Δυτικά Βαλκάνια. Εγώ είμαι συγητή για το Μαυροβούνιο, που τα πράγματα πάνε καλά. Ήμουν εκεί πριν από δύο εβδομάδες και σας συγχαίρω, διότι δημιουργήσατε, ξεκινήσατε τι ομιλίες Σερβίας Κωσυφοπεδίου. Εγώ πάντα υποστήριζα πιο εφάνταστη προσέγγιση για τη διευθέτηση των συνόρων. Δηλαδή, γη για ειρήνη, κάτι όπως γίνεται μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Τα σύνορα του Κωσόβου δεν θα πρέπει να είναι εντελώ άκαμπτα, χωρίς διαπραγμάτευση. Διαφορετικά το κοσυφοπαίδιο για το εκείς μέλλον θα είναι ένα είδος Ταϊβάν στην Ευρώπη. Ο μισός ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει και άλλοι μισοί θα αναγνωρίζουν. Άρα είναι εξαιρετικά βέβαιο το μέλλον και είναι τεράστιο βάρο για του φορολογούμενου μα. 200 εκατομμύρια το χρόνο για τη Γιούλεξ και μόνο. Και υπάρχει α, τεράστιο συνονθήλευμα διεθνών οργανώσεων από την K4, αν και λοιπά που είναι εκεί. Και δεν φαίνεται να υπάρχει μια στρατηγική εξόδου. Είναι πάρα πολύ καλή αυτή που είναι εκεί επί τόπου, κάνουν πάρα πολύ δύσκολη στρατηγική, ε, στατι, ε, πολύ δύσκολη δουλειά. Πώ μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί. Και τι γίνεται όσον αφορά για το καθεστώ οι συνομιλίε μεταξύ Σερβία και Κωσυφοπεδίου που την αιγίδα σα. Ευχαριστώ. Λέζινγκ για τρία λεπτά, κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε, κυρία Άστον, για τη δυνατότητα που μα δίνετε να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων αυτήν από την επικαιρότητα. Θα ήθελα να θίξω την ε, βία στην Δυτική Σαχάρα και να ήθελα να σας ζητήσω να τοποθετηθείτε, κυρία Άστον. Εδώ και εβδομάδες 14.000 ε, έως 20.000 κάτοικοι της Σαχάρας από διαμαρτυρία κατά των Μαροκινών, της Μαροκινής κατοχής, ε, ε, διαμαρτύρονται και καταγγέλουν α, την παράνομη κατάχρηση των φυσικών πόρων στη Βυτική Σαχάρα από τους Μαροκινούς. Αυτό θα έπρεπε να κινήσει την ε, παγκόσμια κοινότητα και την Ευρώπη. Και το προηγούμενο α, Σαββατοκύριακο η βία κορυφώθηκε και η Μαροκινή αστυνομία πυροβόλησε διάφορους ε, α, Επτά τουλάχιστον τραυματίστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει, λέει, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά συνεργάζεται με το Μαρόκο. Στενά. Το οποίο έχει προβεί σε παράνομη κατοχή και οφείλεται σε, στο Μαρόκο η κατάδια των ανθρώπων αυτών. Πώς μπορεί να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει προκειμένου και ο νέος αυτός που χάθηκε από τα πυρά των αστυνομικών να μην ο θάνατός του να μην ε, μείνει ατιμόρυτος. Τι θα κάνουμε, θα γίνουν έρευνες από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βρεθούν οι υπέτειοι και πώς θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση τη μελλοντική συνεργασία με το Μαρόκο. Μία άλλη ερώτηση για την Σομαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια επιχείρηση στη Σομαλία αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί με το TFG, το οποίο όχι μόνο χρησιμοποιεί παιδιά πολεμιστές, αλλά και οφείλεται για εγκλήματα πολέμου. Είναι υπεύθυνη για εγκλήματα πολέμου. Σε παρόμοιες επιχειρήσεις στο παρελθόν, το TFG έχει χρησιμοποιήσει και πολίτες ε, άμαχους. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα σοβαρά και σας ρωτώ πώς αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κυρία Λέζιν. Να δώσουμε ένα περιθώριο στην ύπατη εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο να δώσει απαντήσεις. Έπρεπε να κλείσω τον κατάλογο των ε, αγορητών. Ε, δεν, μπορούμε να... δεν υπάρχει περιθώριο να δεχτούμε κι άλλους. Έχετε το λόγο, Βαρόνι Άστον. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου? 7-8 λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις. Είχα προβλέψει ότι θα ξεπερνούσατε τον κατάλογο με τα θέματα. Σας ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα και εσάς και όλους τους υπόλοιπους για τα ευγενικά σας λόγια, για την Κούβα είναι σημαντικό να δούμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο. Είπαμε στο Συμβούλιο ότι χρειάζεται ένας χρόνος προβληματισμού και στο πλαίσιο της κοινή συμφωνίας. Τίποτα δεν αλλάζει προς το παρόν. Και θα γίνει ένα είδος βολιδοσκόπησης, όπως είπε και ο Γερμανός υπουργό. Δηλαδή, θα αρχίσουμε διακριτικά να εξετάζουμε διάφορα θέματα. Η θέση δεν έχει αλλάξει. Η θέση είναι αμετάβλητη. Και ο Χαβιέρ Σολάνας, ένας από τους προκατόχους μου, είχε πει ότι δεν αρκεί αυτό. Και αυτό αντιλαμβάνεται και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτού του βραβείου, του βραβείου Ζαχάροφ που απονεμήθηκε στον κύριο Φαρίνες και είναι σημαντικό να το παραλάβει και αυτό προσώπος. Πάντως το Συμβούλιο είπε προβληματισμός, μία περίοδος προβληματισμού, τίποτα παραπάνω δεν υπόθηκε. Κύριε Βιγγένιν, σας ευχαριστώ για το σχόλιά σας για τους ε, στρατηγικούς εταίρους. Τώρα, πώς μας επηρεάζουν, πώς ε, αντιλαμβανόμαστε το ρόλο τους. Έχουμε πολλούς στρατηγικούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και είναι πολύ διαφορετική μεταξύ τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τέτοιος εταίρος. Και για τον καθένα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε αντίληψη για τη σχέση που θα έχουμε. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Κίνα, Ινδία. Εκεί βλέπουμε υπερδυνάμεις ή δυνάμει, μεγάλες δυνάμεις που έχουν τη δυνατότητα εξαιτίας των οικονομικών και πολιτικών μας σχέσεων να επηρεάσουν και τη δική μας καθημερινότητα και είναι δυνητικά και ισχυρή εταίροι σε πολλές από τις δικές μας δραστηριότητες. Για το θέμα της πειρατείας, για παράδειγμα, και με την επιχείρηση Αταλάντη. Και συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα. Υπάρχει ένας συνδυασμός δηλαδή μεταξύ των ε, χαρακτηριστικών των διμερών μας σχέσεων και εκεί ερωτώ και τα 27 κράτη-μέλη να σκεφτούν ποιος θα πρέπει να είναι ο πυρήνας και η ουσία αυτών των σχέσεων και πώς θα εξασφαλίσουμε αφίδρομες σχέσεις. Αλλά κάτι τέτοιο προποθέτει μια σαφή και δηλωμένη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα συνδυασμό των οικονομικών σχέσεων και του πολιτικού διαλόγου και της ενότητα μεταξύ μας και του, ναι, της ε, επισήμασης θεμάτων που είναι σημαντικά για μας, όπως είναι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά βλέπουμε και το ρόλο που διαδραματίζουν αυτοί οι στρατηγικοί εταίροι στο παγκόσμιο προσκήνιο, προσκήνιο ή το ρόλο που τους οθούμε να παίξουν. Για το διάλογο και το χρονοδιάγραμμα, επειδή υπευλήθη και από άλλους συναδέλφους, θα το σχολιάσω αργότερα. Κυρία Νέιτ, σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια, τους δύο υψηλόβαθμους διορισμούς. Όντως, είναι πολύ ταλαντούχοι οι δύο συνάδελφοι και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφώνησαν να στελεχώσουν την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και κάτι που θα γίνει όλο και πιο σημαντικό και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για, τα, για τις παγωμένες συγκρούσεις στην υπερδινιστερία. Με το 5 συν 2, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, το συζητήσαμε και με τον Σεργέη Λαυρόφ, τον Ρώσο Ιπέξ, και όταν σκεφτόμαστε και το μέλλον της Μολδαβίας, έχουμε υπόψη και τις παγωμένες συγκρούσεις. Πάντως αυτό είναι κοινό ε, κοινό στόχο του Κοινοβουλίου, ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις παγωμένες συγκρούσεις και με την πρόληψη των συγκρούσεων και με την ανοικοδόμηση της ειρήνης. Για το Αφγανιστάν, εγώ ε, ενδιαφέρομαι κυρίως για τις καλές πολιτικές αποστολές, αστυνομικές αποστολές. Θέλω να είναι ασφαλής ε, το προσωπικό μας εκεί και να μπορέσουν οι δικές μας αποστολές να βοηθήσουν το λαό του Αφγανιστάν. Αυτό είναι αυτό είναι ο δικό μου στόχο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τι επαφέ που είχα, σα μίλησα για την ε, Μέση Ανατολή, Συρία, Ιορδανία, Αραβικό Σύνδεσμο, Αίγυπτο κτλ. Όλοι αυτοί η εντέροι είναι σημαντικοί για να δώσουν όθηση στην ερευνητική διαδικασία. Κύριε Λούνατσεκ, για την ε, ανοικοδόμηση της ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ασχολούμαστε και με τη διαχείριση των κρίσεων και είναι ένα οριζόντιο θέμα σε όλες μας τις δραστηριότητες. Δεν είναι θέμα μιας... Δεν είναι κάτι αποσπασματικό. Αυτό το κάνουμε και στην Ινδία και στο Πακιστάν, σε όλες τις χώρες του κόσμου που δρούμε. Έχουμε 135 αντιπροσωπείες. Πάνω από 100 χώρες δυνητικά θα επηρεαστούν και από τις κλιματικές αλλαγές μόνο. Οπότε μα ενδιαφέρει το θέμα τη ασφάλεια και το τι συμβαίνει στι διάφορε περιοχέ του κόσμου. Και θέλω να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαντικό ρόλο παντού. Τώρα για τη Σερβία, για το κοσυφοπέδιο Το χρονοδιάγραμμα των συνομιλιών ε, έχει τεθεί από τον πρόεδρο Τάντιτς και τον πρωθυπουργό Τάτσι. Το κοσυφοπαίδιο θα γίνει με ήπιο και διακριτικό τρόπο. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των, των αυτών και εκείνα, από εκεί να ξεκινήσουμε την πρόοδο. Τώρα, πόσο θα προχωρήσουμε και τι θα καλύψουμε θα εξαρτηθεί από το πόσο θα καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα το πρωί συζητούσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα των θεωρήσεων και για τον Πρωθυπουργό Τάτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό Έχετε δίκιο ότι το Κωσυφοπέδι είναι μια χώρα που θέλει να προχωρήσει, αλλά έχετε δίκιο και για την ε, ευρωπαϊκή πρόπτικη. Ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να σημειώσει πρόοδος. Ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και το, την πρόταση των Ισραηλινών ή την περιγραφή που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για το κράτος και για τους πολίτες τους. Οι Παλαιστίνοι είπαν ότι αυτά δεν είναι θέματα που θα συζητηθούν τώρα. Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στα πλαίσια ενός ευρύτερου πακέτου που θα διέπει και το καθεστώς όλων των ανθρώπων στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Κύριε Προβέρα, μιλήσατε για τη Σομαλία και είπατε ότι είναι περιτέ οι διεθνεί διασκέψει. Σα διαβεβαιώ ότι πήγα σε μια συνδιάσκεψη που δεν ήταν καθόλου άχρηστη. Συμπροέδρευσα σε αυτήν στο Μαυρίκιο και εκεί ήταν οι Κένια, οι Κομόρες, ε, Μαυρίκιος, πολλές περιφερειακές οργανώσεις, Μοσανβίκη, συμμετείχαν σε αυτή τη διεθνή συνδιάσκεψη και συζητήσαμε για το πώ θα αναπτύξουμε την αφρικανική ηγεσία στον τομέα αυτόν τον αφρικανικό ηγετικό ρόλο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε του Αφρικανού ηγέτε για να ασχοληθούν με ένα ζήτημα που του αφορά άμεσα, του προβληματίζει πολύ και εμεί θέλουμε να του βοηθήσουμε και με του πόρου που χορηγούμε, που είναι δαψιλής, συμφωνώ, αλλά και με το έργο που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και, με, και στη χώρα αυτή. Η προσέγγιση μας είναι συνολική σφαιρική, αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις γειτονικέ χώρες να διαδραματίσουν όσο το δυνατό ισχυρότερο ρόλο. Κύριε Τάνοκ, σας ευχαριστώ για την επιστολή σας το επιτελείο μου, η βοηθή μου ε, το εξετάζουμε πολύ σοβαρά. Φυσικά θέλουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας όλο και πιο αποτελεσματικά και για να εξοικονομήσουμε πόρους όσο γίνεται. Και ένα τμήμα θα επανεπενδυθεί για να ε, εξοικονομηθεί στο μέλλον. Πάντως συμφωνώ μαζί σας. Για το Ανατολικό Σουδάν έχετε απόλυτα δίκιο ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Και όταν ο Μπάνκι Μουν ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξανασυναντηθήκαμε και μας είπε ότι αυτό θα είναι το μείζον θέμα εξωτερικής πολιτικής για τις αρχές του επόμενου έτους. Υποστηρίζουμε και τον πρόεδρο Ταμπέκη, τα θέματα των συνόρων, τα οικονομικά ζητήματα, ζητήματα που δεν καλύπτουν μόνο Βορρά και Νότο. Και οι χώρες του κόλπου έχουν δραστηριότητες στο Νότιο Σουδάν και προσπαθούν να σημειώσουν πρόοδο και ο ΙΕ δραστηριοποιείται εδώ και θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία και ελπίζουμε με αποτελεσματικό τρόπο και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Πάντως όλοι ε, παρατηρούμε με κομμένη την ανάσα τι θα συμβεί εκεί. Και για το θέμα της Unifor ε, μίλησα. Είπατε ότι υπάρχει μια σύγχυση με τις δραστηριότητες μας στα Βαλκάνια. Ελπίζω να μην είναι αυτή η σούπα που περιγράψετε αυτό το, το μπέρδεμα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ελπίζω να γίνει μια ε, διαλεύκανση αυτής της κατάστασης και για το Κωσυφοπέδιο. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Σαχάρα, νομίζω ότι η κυρία Λεφίνγκ, η ειδική επισταλμένη του ΟΗΕ, έχει σημαντικό ρόλο εκεί. Προσπαθεί να ε, παροτρύνει τα συμβαλόμενα μέρη να καθίσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εμείς παρέχουμε και ανθρωπιστική βοήθεια κυρίως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πάντως θα το ξαναελέγξω. Θα, θα ελέγξω τα στοιχεία που δώσατε και εσείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Άστον. Είσαστε ακριβείς όσον αφορά το χρόνο. Δείχνει καλή εκπαίδευση και διανοητική τάξη. Λοιπόν, παρακαλώ, πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο στο 1,5 λεπτό. Αν θέλετε να κάνετε πάνω από μία ερώτηση, κάνετε λιγότερε, μικρότερε παρεμβάσει. Ο πρόεδρο τη Υποεπιτροπή ε, Νταουζόν για την ασφάλεια και την άμυνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπατή Εκπρόσωπο, καταρχά θα ήθελα να σα συγχαρώ για αυτά που κάνατε για την κίνηση του διαλόγου μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Διδραματίσατε κρίσιμο ρόλο στις συζητήσεις με τον πρόεδρο Τάτζης και μπορούμε να σας συγχαρούμε για τα ουσιαστικά αποτελέσματα που πετύχατε. Θα ήθελα να εκφράσω πιο κριτική άποψη όσον αφορά τη σημαντική πολιτική την πολιτική ασφάλεια και κοινή αμήνη που απορρέωνε από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που έχουν κολλήσει πέρα από τι επιχειρήσει που ακολουθούν την δυναμική, την αρχική που είχαν, όπω την Αταλάντα, Αταλάντη που αναφέρατε. Ε, βασική είναι η ευθύνη των κρατών ασχολείται, ασχολείστε πάρα πολύ με τη δημιουργία τη υπηρεσία εξωτερική δράση, αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχει δημοσιονομική χρηματοπιστική κρίση που βαρύνει πολύ σοβαρά τα θέματα τη αμήνη, αλλά τελικά παρόλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες Οι υπουργοί αμήνης εκφράζουν πολλέ ανησυχίε. Είχα, ο κ. Κάμερον δεν αναφέρει την Ευρώπη, τα μιλάει για άμυνα, είδα μια συνέντευξη ε, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αμήνης είναι κάτι θολό. Και όμω μιλάει η Ευρωπαϊκή Άμυνα και μίλησε Ιούλιο και Σεπτέμβριο ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο κ. Ράσμο, με τον οποίο συνεννοείστε πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά αυτά ήταν. Τι πρωτοβουλίε μπορούμε να περιμένουμε από αυτού του θέματος. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε μεγαλύτερη ρόμη σε αυτή την πολιτική, τη νέα και φιλόδοξη στρατηγική που απορρέει και δημιουργείται από την συνθήκη της αγώνας. Ευχαριστώ. Τακτικός και μαζεμένος ο κ. Τανζάν. δούμε αν μπορεί να μιμηθεί ο επόμενος αν ξεκινήσει τα... Α, έφυγε. Παντσέρι, ο κύριος Παντσέρι για 1,5 λεπτό. Ελπίζω και λιγότερο να χρειαστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω που ήρθατε να σας θέσω ένα ερώτημα που ελπίζω να βρει μια απάντηση ικανοποιητική και το θέτω επανειλημμένα μέχρι να βρει απάντηση. Είναι ένα ερώτημα που ήδη το έθεσα πρόσφατα όταν συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι το θέμα των διαφόρων εντολών, των θητιών επίση. Σχετίζεται με τις συμφωνίες πλαίσια με τις άλλες χώρες και σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα παράδειγμα, την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία που θα πάει στη Λιβύη και δεν γνωρίζει αυτή η αντιπροσωπεία την εντολή τι εντολή έδωσε το Συμβούλιο όσον αφορά το δυνατότητα καθορισμού συμφωνίας πλαίσιο. Ζήτησα επανειλημμένα να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Ή είναι ευαίσθητο, απόρριτο το έγγραφο και θα πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο για να μπορέσει κάποιος, κάποιος τρόπος να το συμβουλευτεί αυτό το έγγραφο και αν είναι απόρριτο γιατί και ευαίσθητο. Αν δεν είναι ευαίσθητο και απόρριτο δεν καταλαβαίνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ε, λάβει γνώση αυτού του εγγράφου. Ε, ε, διακυβεύεται και αξιοπιστία του Κοινοβουλίου όταν μεταβαίνει σε άλλες χώρες και αξιοπιστία των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο. Ε, επεξεργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε καλά για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Θα ήταν καλό να κάνουμε κάτι καλό και πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, Αρλάκη, ο κύριο Αρλάκη, για μισή λεπτό. Ναι, ευχαριστώ. Μία μικρή ερώτηση. Μία για το Αφγανιστάν. Δεν πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει μια μεγάλη ευκαιρία για να υποβάλει κάποια σημαντική πρόταση για το θέμα το πρινικό στο Ιράν. Ως τώρα η συζήτηση περιορίζεται μέρα με τη μέρα και τώρα έχει περιοριστεί στο θα επιβληθούν κυρώσεις ή όχι. Δεν πιστεύετε ότι έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της πρότασης Τουρκίας-Βραζιλίας για το ουράνιο της, του Ιράν, το οποίο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί εκτός του Ιράν. Μία πρόταση την οποία αρχικά υποστηρίζαν και το Ιράν και η ΙΠΑ. Και μετά σταδιακά, η οποία πρόταση σταδιακά στη συνέχεια απορρίφθηκε. Εσάς ποια είναι η θέση σας και ποια είναι η θέση σας για την περαιτέρω ε, τον περαιτέρω περιορισμό της συζήτησης. Δεύτερο θέμα, Αφγανιστάν. Βρισκόμαστε στην τελική φάση της της κατάστασης στρατηγικής στο Κοινοβούλιο για το Αφγανιστάν. Ε, εργαζόμαστε επί ένα έτος στα θέματα της στρατηγικής για το Αφγανιστάν και είναι πολύ λεπτομερής η θέση μας. Η στάση της Επιτροπής ως τώρα δεν ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Ελπίζω να παρέμβετε και να διορθώσετε την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Αρλάκη. Ο κύριο Σούλτ, ο πρόεδρο τη ομάδα εργασία, ασχολείται με τη Μέση Ανατολή. Α, συγγνώμη. κύριο Πέτερινγκ, πρόεδρο τη ομάδα εργασία για τη Μέση Ανατολή, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε και Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είσαστε στο καθήκον σα, ε, μάλλον δεν ζηλεύει κανεί. Ε, το καθήκον σας, γιατί έχετε 27 Υπουργού Εξωτερικών και πρέπει να ασχοληθείτε με όλον τον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι σας συνοδεύουμε με συμπάθεια. Αλλά ανησυχούμε και βλέπουμε με μεγάλη ανησυχία κάποιες εξαρτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα στην ομάδα εργασίας για την μέσα Ανατολή. Μέση Ανατολή συζητήσαμε τις δηλώσεις ε, του Αχμαντινετζάντ έναντι του Ισραήλ και θεωρήσαμε φυσικά ότι είναι απαράδεκτε σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ύπαρξη του Ισραήλ. Αλλά επίση λέμε ότι είναι απαράδεκτο και το ερωτώ για το κατά πόσο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο σαφή λόγια, ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίσει το Ισραήλ την πολιτική των απικιών τους. Ούτε η Ανατολική Ισραήλ, ε, η Ανατολική Ιερουσαλήμ ανήκει το Ισραήλ, ούτε μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει τις ε, απικίες στην Ευρωτική Ιορδανία. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ευκαιρία ή δυνατότητα να ασχοληθεί εκ νέου ο ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να σας καλέσω να κάνετε βασική προτεραιότητα της πολιτικής σας στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Ευχαριστώ κύριε Πέτρη και τώρα ο κύριος Μπέρμαν πρόεδρο τη Αντιπροσωπή για τι σχέσει με το Αφγανιστάν. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συμφωνώ με την κυρία Νέιτς, η οποία ανέφερε την ανάγκη να, να, ξανακοιτάξουμε την ευρωπαϊκή πολιτική στο Αφγανιστάν και να επανεξετάσουμε την στρατιωτική μας παρουσία, γιατί η επιτυχία απέχει η παρασάγκας. Μια συγκεκριμένη όμως ερώτηση για τον Αφγανιστάν. Δύο ε, Γάλλοι δημοσιογράφοι έχουν απαχθεί εδώ και 300 μέρες ε, στο Αφγανιστάν και αυτή την εβδομάδα απέχθηκε ένας Ολλανδός δημοσιογράφος. Πότε, πώς θεωρείτε ότι η συνεργασία εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταφέρει να πετύχει την απελευθέρωση των απαχθέντων. Δεύτερη ερώτηση. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Το Wikileaks και σχετική αναφορά για τις καταχρήσεις, τις ευρύτατες καταχρήσεις στο Ιράκ. Έχει ξεκινήσει μία παγκόσμια έρευνα για τον, την κατάσταση. Τι πιστεύετε για την έρευνα αυτή, την υποστηρίζετε? Ευχαριστώ κύριε Μπέρμαν. Κύριος Σούλτς για 90 δευτερόλεπτα. Ναι, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι συχνά έρχεστε σε επαφή και έρχεστε εδώ πέρα στην ε, Επιτροπή μας και έχουμε την ευκαιρία να σας, να σας κάνουμε ερωτήματα για την επικαιρότητα. Το ψήφισμα για την Μολδαβία, το οποίο ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και μια πρωτοβουλία μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, ε, η οποία αναστέλει θέματα με τους πρέσβεις και συνδέεται με το πρόβλημα της υπερνηστερίας. Σας ερωτώ, ποια είναι η θέση σας για την πρόταση αυτή, δραστηριοποιήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση και πώς θα μπορούσε το θέμα αυτό να μην έχει τεθεί στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας που έγινε λίγες μέρες πριν. Ήσασταν ενήμεροι ή συνηθίζετε σε διμερείς συζητήσεις να κάνουν τέτοιες προτάσεις οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Ο κύριος Κέιλαμ, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Άστον που μας εκφράσατε τις ιδέες σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία με την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης πολλές ανησυχίες εκφράστηκαν για ανεπαρκή διατλαντικό συντονισμό και μετά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες ε, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατυπώθηκε ο κίνδυνος ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να φέρει τα κράτη-μέλη αντιμέτωπα μεταξύ τους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμέτωπη με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Συμφωνείτε ότι για να έχουμε πιο εκτεταμένη συνεργασία με τη Ρωσία θα πρέπει προηγουμένω να σεβαστεί οι υποχρεώσεις της ανηλυμένες όπως την εκεχηρία με τη Γεωργία. Την επόμενη φορά που θα συναντηθείτε με τους ομολόγους σας από τη Ρωσία μπορείτε να εκφράσετε, να διαβιβάσετε την ανησυχία των ε, Ευρωπαίων βουλευτών για την ε, εικονική δίκη ουσιαστικά που έγινε πρόσφατα και που δείχνει την ε, αστάθεια του ρωσικού δικαστικού συστήματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρντεν κλείνει αυτό το κύκλο των παρεμβάσεων για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, καλησπέρα, Βαρόνι Άστον. Δεν περισσεύει ο χρόνος και θα εστιαστώ σε ένα θέμα. Το θέμα της Ζιμπαμπούε, το οποίο δεν νομίζω ότι ετέθη σήμερα το απόγευμα. Αυτό που ανησυχεί όλος ιδιαίτερος είναι η μονομερής διορισμός από τον Μουγκάμπε πρεσβευτών κυρίως διορισμός πρεσβευτού της κυρίας Μουτσάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, αυτό, με αυτό δεν συμφώνησε ο Πρωθυπουργός του Ζιμπάμπου, είναι οι άνθρωποι του Μουγκάμπε που διορίζουν πρεσβευτές και ο Τσαγκαράι ο ίδιος ήρθε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε ότι τα διαπιστευτήρια της θα πρέπει να απορριφθούν. Ποια είναι η διαδικασία. Τα διαπιστευτήρια υποβάλλονται στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου έστειλα και στους δύο επιστολή, και στον κύριο Μπαρόσο και στον κύριο Βαν Ρόμποϊ, στον πρόεδρο του Συμβουλίου, δοθέντος του ρόλου σας στους τομεί και την δυτή σα ιδιότητα, φαντάζομαι ότι έχετε κάποια επιρροή επί του θέματος και θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση να υποστηρίξετε την ιδέα, τα διαπιστευτήρια της κυρίας Μουτζάντα και οδήποτε άλλου πρεσβευτού που έχει διοριστεί μονομερός από τη Ζιμπάμπουε να απορριφθούν. Αυτό θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ κύριε Βανόρντεν. Το λόγο τον έχει βαρώνει Άστον Ξέρουμε την τάξη της σκέψης σας και την παιδεία σας, λοιπόν παρακαλώ αν μπορείτε να τηρήσετε το δεκάλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να το κάνω, σας κάνω τη χάρη. Κύριε Ντονζό, σας ευχαριστώ για τα σχόλια, για το κοσυφοπαίδιο. Τα θέματα ασφαλείας και αμήνης τα βλέπω διαφορετικά. Γευμάτισα με τους 27 επικεφαλείς ε, των, των Υπουργείων Άμυνας των Γενικών Επιτελείων, της επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων και συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα. Ε, είναι ένα θέμα της απασχολείως ιδιαίτερω. Πρέπει όταν εξετάζουμε θετικά θέματα να έχουμε το σωστό πλαίσιο. Δηλαδή πώς στατηγικά συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια μέσα χρησιμοποιούμε για να αντιμετωπίσουμε διάφορα υποβόσκοντα ε, θέματα και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε σωστά στις δομές που έχουμε τα διάφορα ζητήματα που σας δημιουργούν προβληματισμό. Έχουμε καλύτερο έλεγχο των πραγμάτων από ό,τι θεωρείτε. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του κ. Κάμερον. Σε πολλά κράτη-μέλη θα δείτε ότι οι πρωθυπουργοί ε, ε, ε, εξετάζουν τα θέματα μήνυς στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας κλπ. Και γι' αυτό χρειάζεται σωστή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα ε, βλέπω διάφορους ανθρώπους σε συνεντεύξει για τον επικεφαλή της υπηρεσία και ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να μπορούν να προσφέρουν προς τη θέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέποντας και αναγνωρίζοντα ότι σε περίοδο οικονομική ύφεση όταν οι προπολογισμοί είναι σφιχτοί δεν μπορούμε να προσφέρουμε πολλά για την καινοτομία και την έρευνα. Χρειάζεται μια προσέγγιση που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν βέβαια τι αμυντικέ του ικανότητε, αλλά να υπάρχει αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Όταν συναντώνται η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συναντηθούν, θα το συζητήσουν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ συναντώμε τακτικά με το Γενικό Γραμματέα Ράσμουσεν. Συζητούμε τη μεγαλύτερη συνεργασία, συντονισμό, ούτω ώστε τα πολιτικά ζητήματα να μην επηρεάζουν τη δυνατότητα συνεργασίας μας επί τόπου. Και με τον στρατηγό Πατρέας ε, συναντήθηκα περασμένη εβδομάδα, συζητήσαμε τι κάνουμε στο Αφγανιστάν και πόσο αποτελεσματική συνεργασία είναι εκεί. Είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μου. Σωστά τα είπατε. Υπάρχουν και περισσότερα πρέπει να γίνουν και είναι ένας τομέας που ήδη συζήτησα με το γενικό γραμματέα που θα αναλάβει σε λίγο, το γενικό μας γραμματέα που θα αναλάβει τα καθηγοντά σε μερικές εβδομάδες ότι πρέπει να εστιαστεί σε αυτά τα θέματα. Κύριε Παντζέρη, θέσατε ένα ζήτημα. Ξέρω την απογοήτευσή σα, Τα άκουσα στη φωνή σα πόσο απογοητευμένος είστε και πόσο ανησυχείτε. Ποια είναι η δυσκολία, ότι δεν έχω μόνη μου στα χέρια μου αυτό το θέμα, δεν μπορώ να το λύσω μόνο μου. Πρέπει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονιστούν και θα διεξαχθούν συζητήσει στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων την επόμενη εβδομάδα και εκεί θα συμβάλλουμε συζητήσει Εγώ έχω στόχο την ταχύτερη δυνατή λύση, δεν μπορώ να προβλέψω πότε, αλλά καταλαβαίνω την ανησυχία σας κυρίως όταν ταξιδεύετε και φέρετε αποτελέσματα. Θα διαβιβάσω την απογοήτευσή σας και είδα που κι άλλοι κούναγαν το κεφάλι τους όταν εκφράζατε τις ανησυχίες σας και σας καταλαβαίνουν. Να στραφώ τώρα στο θέμα του Αφγανιστάν και τα σχετικά σχόλια και ερωτήσεις. Κάπου έβαλα τη σελίδα μου. Έχασα τη σελίδα μου δυστυχώς. Λοιπόν, να μιλήσω για το Αφγανιστάν να ψάχνω για τη σελίδα. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι έγινε καλή προσπάθεια εκεί. Δεν ξέρω τι εννοούσατε όταν είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εφαρμόζει αυτά που είπε. Ρωτήσατε για το Ιράν. Βρήκα το χαρτί μου. Αν χάνουμε την ευκαιρία. Μήπως δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντά μας. Αν δεν εξετάζουμε διάφορες προσεγγίσεις. Κοιτάξτε, προσπαθούμε. Προσπάθησα να ξεκινήσω τις συζητήσεις, ανέλαβα πρωτοβουλίες, δεν τις περιγράψω. Χρειάζεται ξεκάθαρη προσέγγιση. Οι συζητήσεις μας με το Ιράν αφορούν τα θέματα πυρηνικής ικανότητας και όχι άλλα θέματα. Αυτό εκεί πρέπει και θέλουμε να είναι άκρως επικοδομητικές οι συνομιλίες. Συζήτησα για το θέμα της πρωτοβουλίας της Τουρκίας και της Βραζιλίας για το Ιράν με του Είναι ξεχωριστό ζήτημα αυτό. Ξεχωριστό από αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή, ποιο είναι το πυρηνικό δυναμικό του Ιράν Υπάρχουν και άλλα παράλληλα θέματα, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό το βασικό θέμα. Κύριε Πέτερινγκ. Μιλήσατε για, το, για τις δηλώσεις για τα όσα είπε. Ελπίζω να ακούσατε τα σχόλια που έκανα και τι προσπάθησα να εκφράσω για το θέμα των επικισμών ήμουν ξεκάθαρη όσον αφορά τους επικισμούς. Ο ΙΕ θα πρέπει να συμμετάσχει περισσότερο. Το θέμα είναι κατά πόσο οι συνομιλίες μπορούν να ξαναξεκινήσουν. Οι ΙΠΑ μπορούν να φέρουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με κάποιο ψήφισμα για το μορατόριουμ και να μην οδηγήσει μετά από ένα-δύο μήνες άλλο εμπόδιο, αλλά να βρούμε μια δέξοδο. Το κουαρτέτο το υποστηρίζει αυτό. Συνεργαστήκαμε, συνομιλήσαμε, κινούμεθα ενεργώς. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τη διαδικασία. Είναι τεράστια προτεραιότητα για μας. Πήγα τρεις φορές στη Μέση Ανατολή φέτος. Το συζήτησε επανειλημμένα. Το έχουμε σαν προτεραιότητα ύψιστη. Και όσο προχωρούν οι συνομιλίες θα υπάρξει περιθώριο να κάνουμε περισσότερα. Κύριε Μπέρμαν, δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που ε, συμβαίνουν στον αφορά την απαγωγή. Καταλαβαίνω τα συναισθήματά σας. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει τους υπηκούς της σε περιοχές όπως είναι το Αφγανιστάν. Αυτό το συζητάμε και να προσφέρουμε όποτε ενδείκνεται υποστήριξη και στα κράτη-μέλη και όποτε χρειάζεται το κάνουμε σας διαβεβαιώνω. Κύριε Σούλτς, Μολδαβία αν γνώριζα, αν αναμίχθηκα, αν ήξερα τα όσα υπόθηκαν με την καγκελάριο Μέρκελ και τη συζήτηση με τη Ρωσία, ναι, είναι σημαντική αυτή η διμερής διάλογη, αλλά υπάρχει τεράστιος όγκος επικοινωνιών που λαμβάνει η χώρα συνεχώς μεταξύ ημών με Ήτα και των κρατών μελών και συμμετέχουμε. Δίκιο έχετε. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον, οι μελλοντικέ σχέσει με τη Μολδαβία και τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την υπερδνηστερία. Κύριε Κάλαν, υπερατλαντικό, διατλαντικός συντονισμός, σημαντικότατος, συμφωνώ. Αυτό που είπατε, ότι η Ρωσία θα πρέπει να τηρήσει τις πρώτερε υποχρεώσεις. Δεν ξέρω αν ανέλαβαν αυτή την υποχρέωση σαν τις που ήλπιζα και ευχόμουν να αναλάβουν. Πάντα θέτουμε τα θέματα αυτά, τις ανησυχίες που εκφράσατε για τα άτομα, για τις εικονικές δίκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη γεωργία, πάντα είναι στην ημερήσια ένταξη των συζητήσεων. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να δημιουργήσουμε καλή εταιρική, συνεργασία, εταιρική σχέση με τη Ρωσία, όπου καλύπτονται, συζητούνται αυτά τα θέματα. Να μπορούμε να προχωρούμε στην εταιρική σχέση για τον εξυγχρονισμό, και έτσι μπορούμε να πετύχουμε την οικονομική συνεργασία που θέλουμε και τη θεσμική συνεργασία. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και αυτό κάνουμε. Τέλος. Κύριε Βανόρντεμ, είχατε την καλοσύνη να με να με ενημερώσετε σχετικά με την επιστολή που στείλατε στους δύο προέδρους. Είναι πολύ ενσυχητικό αυτό. Δεν ξέρω που θα καταλήξει η συζήτηση με τους Προέδρους, αλλά άκουσα αυτό που είπατε. Αν θέλουμε να έχουμε έναν πρεσβευτή, θα πρέπει να μιλάει εκ μέρους της χώρας του, της χώρας που εκπροσωπεί. Και οι δύο Πρόεδροι το συζητούν το θέμα. Θα κινηθώ ξεχωριστά, ξέρω περισσότερο ποιες είναι οι σκέψεις τους και θα σας ενημερώσω δεόντως. Σας ευχαριστώ Βαρόνι. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Χάουταλε, κυρία αλλά πρόεδρος της Υποπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 1,5 λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα θερμά να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος Παντσέρη για την ανεπάρκεια και την ε, ανεπαρκή πρόσβαση των ε, σωμάτων ε, του Κοινοβουλίου σε τέτοια βασικά στοιχεία για τις εργασίες μας. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα αποτελέσματα ε, των εταιρικών σχέσεων με την Κίνα, με τη Ρωσία, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μία θέση με σύγχυση. Κοιτώντα τι έγινε στις 6 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι είναι κοινή νοήματος ε, η σύνοδος και χωρίς κανένα αποτέλεσμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόσφατα ε, ο κόσμος ξύπνησε για κάνα δύο μέρες με την απονομή του βραβείου Ειρήνης Νόμπελ. Ποια είναι η στρατηγική σας στο σημείο αυτό. Να σας θυμίσω κατά τρίτον ότι Εξ ονόματος της Επιτροπής μας ε, σας αποστήλαμε μία επιστολή γιατί ανησυχούμε ότι μπορεί να μην θυμόσαστε για ότι δεν μπορεί να θυμόσαστε τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει για τις δομές σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό στο, στο έργο. Ευχαριστώ κυρία Χαρτ αλλά η κυρία Γιαννάκου για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ύπατη εκπρόσωπο για την παρουσία της εδώ. Έχω τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ε, κυρία εκπρόσωπε, ποιος θα είναι ο ρόλος της συμμετοχή των Ρώσων στο Αφγανιστάν. Δεύτερον, στην επικείμενη συνάντηση Ευρωπαϊ... Ανώτατη ε, Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών θα συζητηθεί το θέμα Wikileaks. Και τρίτον, έχετε ήδη αποφασίσει για, την, ε, για το European Defense Agency για το ποιον θα τοποθετήσετε γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιαννάκου. Κυρία Μποσκούρ για μισή λεπτό. Ναι, λυπάμαι, δεν ακούστηκε το όνομά μου. Μία ερώτηση έχω να κάνω για την Κίνα και συμφωνώ ναι. με την κυρία Ουτάλα. Θα ήθελα να προσθέσω το θέμα των Ουιγούρων στα ανατολικό τμήμα της Κίνας, οι οποίοι πλήττονται καθότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται και δεν έχουν επαφή με ακόμα και γιατρούς στις φυλακές. Δεύτερη ερώτηση για την Τουρκία. Από τότε που εσείς ε, πήγατε με τον κύριο Φιούλε τον Ιούλιο στην Τουρκία, ξεκίνησε και στρατηγικός διάλογος. Μία ερώτηση λοιπόν που έχω να σας κάνω είναι η εξής. Ε, είναι σημαντικό το θέμα του διαλόγου, αλλά φυσικά παντού ανακύπτει το θέμα της Κύπρου. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να βοηθήσετε όλες τις πλευρές να προωθήσουν μία λύση την οποία χρειαζόμαστε όχι μόνο για την ίδια την Κύπρο, αλλά και για τις σχέσεις με την Τουρκία και την όλη διαδικασία της Τουρκίας. Σας ευχαριστώ κυρία Μποσκούρ. Σάκε για 1,5 λεπτό. Κυρία Σάκε. Ευχαριστώ Πρόεδρα και είπατε εκπρόσωπα. Το πακέτο για τις κυρώσεις για το Ιράν ε, πρόσφατα ε, επικυρώθηκε για το Ιράν. Και αναφέραμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι στοχοθετημένες οι κυρώσεις για το Ιράν αν είναι στοχοθετημένες οι κυρώσεις, θα πρέπει να έχουν και κάποια ακρίβεια, την οποία αναφέρατε και στην προηγούμενη απάντηση που δώσατε. Τώρα μάθαμε ότι έχουν αποσταλεί φορτία μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να τα αντιληφθούμε και ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ασκήσει πίεση στις ενεργειακές εταιρείε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουν συμφωνίες σε ό,τι αφορά και το Ιράν. Πέρα από τις ε, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, για παράδειγμα, έχει οδηγήσει στον περιορισμό των ανεφοδιασμού στο Ιράν με βρετανικών αεροσκαφών και εκ παραλίλου αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να επηρεάζονται οι ροές πετρελαίου και αερίου και προς το Ιράν. Ποια είναι η αντίδρασή σας στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα θέσετε στην επόμενη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα και παρά το γεγονός ότι έχω εκφράσει αμφιβολίες για τις κυρώσεις, θεωρώ ότι οι κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να επιφέρουν αποτελέσματα. Θα τα εξετάσετε αυτά. Σας ευχαριστώ κυρία Σάκη. Στράσερ για μισή λεπτό. Ο κύριος Στράσερ. Ευχαριστώ την ε, είπατε εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ για τα σαφή λόγια που χρησιμοποιήσατε, όχι μόνο στην εισαγωγή σας, αλλά και στις απαντήσεις σας. Θεωρώ ότι είναι καλή η συνεργασία με την Επιτροπή και θα ήθελα να υποστηρίξω τον συνάδελφο Παντσέρη σε ό,τι αφορά τη Λιβύη. Θα θέλαμε και εμείς τις απαραίτητες πληροφορίες και σίγουρα η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το θέμα με την κατάλληλη εμπιστευτικότητα. Να συζητήσω και εγώ την 20η Νοεμβρίου την Σύνοδο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα ΕΕ. υπό την ιδιότητά μου ως ε, σκιώδης εισηγητής για το SWIFT τότε και ως ε, εισηγητής για το PNA θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα θέματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των πολιτικών ε, δικαιωμάτων το θέσατε στο επίκεντρο των συζητήσεων με τη ΣΥΠΑ, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά το SWIFT, το PNA, η Συμφωνία γενικότερα για την προστασία των δεδομένων και ακούμε τώρα ότι προγραμματίζεται η κατάρτιση νέας νομοθεσίας στη ΣΥΠΑ και πολλά τέτοια παρόμοια θέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση γενικότερα των θεμάτων αυτών και προς αυτήν την κατεύθυνση χρειαζόμαστε και τη δική σας ε, συνεισφορά. Ευχαριστώ κύριε Στράσερ και τώρα ο κύριος Τάλερ. 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν παρακολούθησα από την αρχή την παρουσίαση και τη συζήτηση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΟΗΕ. Ποια είναι η στρατηγική σας? Πώς πιστεύετε ότι θα είναι πιο επιτυχής ε, η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την διπλωματική σας επιτυχία ε, με τον πρόεδρο Τάντιτς και το κοινό ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το κοσυφοπαίδιο. Θα σας παρακαλούσα να χρησιμοποιήσετε το κύρο σας και να επιμείνετε ώστε να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαπραγματεύσεις ε, με τη Σερβία. Καμία κυβερνητική κρίση, καμία εκλογική κρίση δεν πρέπει να δημιουργήσουν πρόσκομα στην έναρξη των διαπραγματεύσεων και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι μπορείτε να συμβάλλετε τα μάλα. Ας μην ξεχνούμε και τη Μακεδονία. Η κατάσταση στη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, είναι πολύ κακή, πολύ δεινή και ίσως εκεί υπάρχει μια λανθάνουσα σύγκρουση που μπορεί να εξουδετερώσει όλες μας τις επιτυχίες και τα επιτεύγματα στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα παρακαλώ να αναμειχθείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Τάλερ. Κάμπελ για 1,5 λεπτό. Κύριος Κάμπελ. Βαρόνι Άστον, διορίσατε τον πρώτο πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο πρώτος από πολλούς πρεσβευτές που θα αναλάβουν τις θέσεις τους σε πολλές χώρες και θα υποστηριχθούν από 7.000 εκπροβευμένους υπαλλήλου τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αυτό παρεμποδίζει εθνικέ πρεσβείες κατά την άποψή μα. Εγώ σας θέτω. Ο πραγματικός λόγος για την μη αναγκαία αυτή επικάλυψη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει το τέταρτο η τελευταίο στοιχείο ενός κράτους έθνους υπό τους όρους της συμβάσεως του Μοντεβιδέο. Δηλαδή να ξεκινά και να ασκεί διπλωματικέ σχέσεις. Αρνείστε ότι η δουλειά σας κινητοποιείται από, επιθυμία να καλύψετε τα κριτήρια της συμβάσεως του Μοντεβιδέο και έτσι να επιτρέψετε τη δημιουργία ενό κράτου που θα ονομάζεται Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κλείνει το γύρο των παρεμβάσεων. Κυρία Γιάτεμάκη με 1,5 λεπτό. Σα Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την είπατε εκπρόσωπο για την επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι τώρα στα καθήκοντά της. Σε ό,τι αφορά το Αφγανιστάν και την πολιτική στο Αφγανιστάν. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές, τις μη στρατιωτικές προσπάθειες και τις αστυνομικές επιχειρήσεις. Είναι αρκετές οι ικανότητες ε, επαρκής ο μηχανισμός ή χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις και θα πρέπει να στείλουν περισσότερες δυνάμεις στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν φύγουμε, πριν εγκαταλείψουμε το Αφγανιστάν και ίσως και κάποιες ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα, αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχετε εσείς, είπατε εκπρόσωπε, για 10 λεπτά. Thank um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Χάουταλα, και εσείς εκφράσετε την επιθυμία διεξοδικής ενημέρωσης. Το μήνυμα ελήφθηκε από τον κύριο Παντσέρη προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις. Στην ε, διάσκεψη κορυφή με την Κίνα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν στο πρόγραμμα, ήταν στην ημερήσια διάταξη και είναι στα προγράμματα όλων των, όλων των συναντήσεων και των δικών μου όποτε πηγαίνω στην Κίνα. Πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο πρόγραμμα των συζητήσεων. Και ένας από τους λόγους που προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τις δραστηριότητες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, από πλευρά των θεσμικών οργάνων είναι για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μα. Μερικέ φορέ είναι σημαντικό να έχουμε ξεχωριστού και σαφεί διαλόγου με του διάφορου εταίρου μα για τα θέματα αυτά. Άλλε φορέ όμω θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι κεντρικό τμήμα του γενικότερου διαλόγου. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να παραγωνίζονται πάντω ή να περιθωριοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να αποτελούν απόσπαστο τμήμα όλων μα των δραστηριοτήτων. Και αυτή είναι η δεδηλωμένη επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποφασιστικότητα να προωθήσουμε αυτό το σημείο. Και φυσικά δεν θέλουμε απλώς να χανόμαστε σε μεγαλεπίβολες δηλώσεις και σε ρητορική. Μας ενδιαφέρουν τα απτά αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για το έργο το δικό μου στο μέλλον φυσικά από την άποψη ενδιαφερόμαστε και για τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Γιαννάκου, πραγματικά μερικέ φορέ δεν μπορώ να προφέρω τα ονόματα, σα ζητώ συγγνώμη, είμαι ανεπίδεκτη στην προφορά. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, θα... δεν ξέρω ακόμη ποιο είναι επικεφαλής, μόλις ενημερωθώ, ε, θα γίνει αυτή την εβδομάδα, θα σας ενημερώσω άμεσα. Επίσης, ε, θα πρέπει να διοριστεί και ο αναπληρωτή Γενικός Διευθυντής, ε, μετά την, το διορισμό του Γενικού Διευθυντήου θα οριστεί, και ο αναπληρωτής. Για το Wikileaks δεν πρόκειται να κάνω δηλώσεις. θα ακούσαμε μεγάλη προσοχή αυτά που λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα ήταν αδόκιμο να προβώ σε σχόλια. Μέχρι στιγμή δεν ήταν τμήμα του διαλόγου που είχαμε τι Πολιτείε. Κυρία Μποσκούρτ, με ρωτήσατε για την Τουρκία και την Κύπρο. Εγώ δεν συμμετέχω στις συζητήσεις για την Κύπρο ως κράτους μέλους. Οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούν να επιλύσουν το πολιτικό ζήτημα. Πάντως, εγώ παρακολουθώ ενεργά τις συζητήσεις με την Κύπρο ως κράτους μέλους για θέματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο, στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και από αυτήν την άποψη έχω συνεχείς επαφές. Υπάρχουν κάποιοι ρεαλιστικοί τρόποι που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα για να βελτιώσουμε την κατάσταση επιτόπου και υπάρχουν και τα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Και στις συζητήσεις και επαφές που έχουμε με την Τουρκία, ιδιαίτερα τον Τούρκο ΙΠΕΞ, εγώ με σαφήνεια είπα ότι θέλω να καταλήξουμε σε, μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος που θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε τη σελίδα και να δώσουν μια απάντηση στο λαό της Κύπρου. Κυρία Σάκε, για το Ιράν, τις κυρώσεις και τις επιπτώσεις τους στον Ιρανικό λαό. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εφαρμόσουμε στοχοθετημένες κυρώσεις. Κυρώσεις που θα βάλλονται κατά των επιχειρήσεων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να ασκηθεί πίεση στο Ιράν για να καθίσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κυρώσεων, αυτό φυσικά είναι μια κρεμότητα και ο στόχος των κυρώσεων σε ό,τι αφορά τις οικονομικές κυρώσεις είναι σαφέστατος είναι τμήμα τη δυτή αυτής προσέγγισης προκειμένου να προωθήσουμε τις συνομιλίε και να καταλήξουμε σε μια διευθέτηση που θα δημιουργήσουν μια ασφάλεια και για το λαό του Ιράν αλλά και για τους λαούς των γειτονικών χωρών και της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ κύριε Στράσε για τα σχόλιά σας ως προς την σαφήνεια των ε, απαντήσεών μου. Έχω βελτιωθεί, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα βελτιωθώ ακόμη περισσότερο. SWIFT, προστασία δεδομένων και δικαιώματα των πολιτών. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το έχουμε συζητήσει και είναι σημαντικό όχι μόνο το θέμα της συμφωνίας, αλλά το να καταλάβει ε, να καταλάβουν οι Ηνωμένες ε, τη γνώμη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου συναντήσεις και θα προγραμματίσουμε συζητήσεις όχι μόνο εδώ αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί ακούσαμε και τους ε, Αμερικανούς ε, κοινοβουλευτικούς και νομίζω ότι είναι σημαντικό το κοινοβούλιο να συμμετέχει στη, στο διάλογο και να δούμε με ποιους τρόπους θα βρούμε αυτές τις πληροφορίες και να εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τη σημασία αυτών των συμφωνιών. Τώρα αν έχετε και άλλες προτάσεις, γιατί παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, μπορείτε να τις υποβάλλετε γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις και φυσικά θα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επαφή γι' αυτό. Κύριε Τάλερ, Ηνωμένα Έθνη, Ανάγκες και Απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς τον ΟΗΕ, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να περάσουμε ψηφίσματα που θα μας δώσουν ε, μια σωστή φωνή στα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρχε ένα πρόβλημα πριν την συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά τη Λισαβόνα θέλουμε να ακούγεται η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπως της αξίζει, γιατί είμαστε και ο σημαντικότερος δωρητής, ε, συμμετέχουμε στις δραστηριότητες και οι επιχειρήσει του ΙΕ. Είμαστε ενεργοί παντού στον κόσμο και είναι λογικό να μπορούμε να θέλουμε να προτάσουμε μια συνολική προσέγγιση και ενιαία εκ μέρου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω να το καταλαβαίνουν αυτό οι χώρες που ζητούν τη βοήθειά μα. Και αυτό είναι ο στόχο μα για την παρουσία μας στον ΟΗΕ. Φυσικά έχουμε συνεχώς επαφές με τον ΟΗΕ Πολλέ φορέ έχω συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μπαν Κιμούν, και συζητούμε για θέματα στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Και με συνεργάτε του ε, συναντιέμαι πολύ συχνά. σα ευχαριστώ για το σχόλιο για τη Σερβία. Πάντως, τα συγχαρητήρια αξίζουν περισσότερο στον κύριο Τάντιτ, τον Σέρβο Πρόεδρο. Οι συζητήσεις ε, θα αρχίσουν σύντομα. Ο κύριος Κουπέριτα στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα μετέβη και η κυρία Χίλαρη Κλίντον. Έγινε επικοδομητικός διάλογος και βλέπω, διαβλέπω ταχείες εξέλιξεις. Θα πρέπει να βρεθεί ισορροπία βέβαια και να αντιληφθεί η Σερβία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι αφοσιωμένη σε όλες τις πτυχές των σχέσεων μαζί της. Όπως σας είπα θα γίνει διακριτική ε, παρουσία αλλά σταθερή. Σε ό,τι αφορά τη ΦΥΡΟΜ είχαμε συζητήσεις ε, και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες με την Ελλάδα, αλλά ελπίζω ότι και εκεί θα σημειωθεί πρόοδο σύντομα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είπα στον, ε, στον Πρωθυπουργό ότι το, η διαθέτηση αυτού του ζητήματος θα τους πάει ακόμη πιο μακριά γιατί έχουν φυσικά ευρωπαϊκή προοπτική. Κύριε Κάμπελ, δεν ε, σωστή αυτή χρήση των πόρων. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τις προηγούμενες ευθύνες μου, όταν συνάπτουμε μια εμπορική συμφωνία εκ μέρους 27 χωρών και 27 χώρες ε, εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία απώλεια δυνάμεων ικανοτήτων ε, των χωρών για θέματα που ενδιαφέρουν τι επιχειρήσει του. Αυτό όμω που μα ενδιαφέρει είναι μια καλύτερη συμφωνία, γιατί όταν έχουμε μία ενιαία φωνή και εκπροσωπούμε 27 χώρε, είμαστε και πολύ πιο ισχυροί στι διαπραγματεύσει. Και σε ορισμένε περιπτώσει, ε, όταν κάποιο εκπροσωπεί 27 χώρε, ε, έχει και μεγαλύτερο ειδικό βάρο. Και στην ε, ειρηνευτική διαδικασία τη Μέση Ανατολή, αυτή η ενιαία φωνή μα επέτρεψε να έχουμε περισσότερο ειδικό βάρο, να γίνουμε πιο δυναμικός κινητήριο μοχλός και να προωθήσουμε τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερούμε από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δράσουν ή του αφαιρούμε αρμοδιότητες. Απλώς ενισχύουμε με, την, με το συντονισμό αυτό την παρουσία μας. Κυρία Γιατενμάκη, αστυνομική αποστολή, αστυνομικέ αποστολές στο Αφγανιστάν και χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από τη χώρα αυτή. Νομίζω ότι είναι καλέ οι αποστολέ μα στο Αφγανιστάν. Είμαστε σαφείς ως προς τους στόχους μας. Τους ε, συνδέουμε και με το έργο μα αλλού. Το συζήτησα με το στρατικό Πετρέους. Νομίζω ότι είχαμε σημαντικά επιτεύγματα και προσπαθούμε να χαράξουμε και την μελλοντική μας πολιτική. Και νομίζω ότι η ηγεσία εκεί έχει, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Πάντως, ε, τις επόμενες εβδομάδες ε, πιστεύω ότι θα έχουμε εντατικοποίηση των προσπαθειών. Σα ευχαριστώ, είπατε εκπρόσωπε. Τελευταίο γύρος των ερωτήσεων ξεκινά από τον πρόεδρο τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Μασρέκ, ο κύριος Νταβίτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βαρόνι Άστον. Και για μένα είστε υπουργό Εξωτερικών και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις δεξοδικές απαντήσεις που είναι όλο και πιο ευρυθείς και να σας ε, πω ότι μερικές από τις κριτικές ή ακόμη και επικρίσεις που σας απευθύνουμε ακόμη και εγώ δεν είναι προσωπικές ε, απέναντί σας αλλά θέλουμε να τις διαβιβάσετε στις ε, χώρες μέλη. Σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς της Συμφωνία είδηση με την Ιορδανία. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Έχετε την πρόθεση να λάβετε θέση για την θανατική καταδίκη εις βάρος του Ταρέκα Ζής που εκδόθηκε χθες. Δεν νομίζω ότι είμαι αφελής όταν λέω ότι ο Ταρέκα Ζής ήταν στην κυβέρνηση του Σαντάμ Χουσέιν. Αυτό που, ήταν, που έλεγε ο Λένιν ο χρήσιμος ηλίθιος και νομίζω ότι στα πλαίσια των αξιών που χαρακτηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να υψώσουμε τη φωνή μας. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, έχετε την πρόθεση, κυρία είπατε εκπρόσωπη, να διορίσετε τους πέντε πρέσβεις στις χώρες που δεν έχουμε ακόμη πρέσβεις. Και τελευταία ερώτηση, φαντάζομαι δεν θα μου δώσετε απάντηση, κάτι αντίστοιχο που συνέβη και με τον κύριο Παντζέρη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τη Δευτέρα βγω για το Λίβανο και χρειάζομαι μια θέση για την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά το ειδικό δικαστήριο για το Λίβανο. Σας ευχαριστώ κύριε Νταβίδ. Νόιζερ είναι το επόμενο όνομα. Κύριος Νόιζερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Υπατέη, εκπρόσωπε. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ Υπουργό Εξωτερικό σας θεωρώ. Γιατί νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δράσουμε συγκεκριμένα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην Βυτική Σαχάρα, στη σύγκρουση με το Μαρόκο. Όχι μόνο επειδή είναι επίκαιρο το πρόβλημα, αλλά επειδή θεωρώ επίσης ότι επί δεκαετίες η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί ε, την ε, σύγκρουση αυτή και δραστηριοποιείται μόνο εφόσον υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα. Είπατε μόλις ότι η Ευρώπη ε, δίνει ανθρωπιστική βοήθεια και κατά τα άλλα ε, ενισχύονται και τα Ηνωμένα Έθνη. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή κοινότητα θα πρέπει να αναλάβουμε πιο μεγάλες ευθύνες, γιατί αυτή η σύγκρουση είναι δίπλα, έξω από τα σύνορά μας και ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Θέλει επιτέλους δουλειά, θέλει επιτέλους κάπου να μείνει, θέλει κάποια στιγμή να συμμετάσχει, να έχει ε, μερίδιο από τις πρώτες ύλες. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει πιο έντονα, να μην πει απλά ότι δίνει ανθρωπιστική βοήθεια. Πώς λοιπόν να δραστηριοποιηθείτε πιο έντονα για να αμβλύνετε την κρίση της σύγκρουσης στο σημείο αυτό. Σας ευχαριστώ. Πέτερλε, για να είστε το κύριο Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί, Λέντι, Άστον, είπατε εκπρόσωπε, Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου. Έχω σπουδάσει ιστορία και γεωγραφία, αλλά έχω την εντύπωση ότι εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερες γνώσεις από ότι εγώ, ωστόσο δεν έχουμε καλύψει ακόμα το σύνολο του χάρτη. Μία ερώτηση λοιπόν για την Κεντρική Ασία. Μας ανησυχεί ακόμα η κατάσταση στο Κυργιστάν. Και φυσικά οι νέες τάσεις που διαγράφονται στο Τζικιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ειδικό απεσταλμένο, τον κύριο Μορέλο, εξαιρετικό. Ωστόσο δεν έχει από μόνος του αρκετή πολιτική βούληση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο σκοπεύετε να πάρετε περαιτέρω μέτρα στην Κεντρική Ασία δεδομένων των τάσεων αυτών, των τάσεων αυτών. Ε, μπορείτε να φανταστείτε ότι θα υπάρχουν νέε εξελίξει και ποιο θεωρείτε ότι θα είναι ο ρόλο τη Ρωσία, γιατί πρόκειται για στρατηγική εταιρική σχέση. Ευχαριστώ, κύριε Πέτερλε, και τώρα ο λόγο τον Σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Με μεγάλη χαρά σας ακούω. Αλλά πρέπει να πω ότι τελικά δεν, έλαβα, δεν άκουσα αυτό που ήθελα όσον αφορά το θέμα του Αφγανιστάν. Συγκρούσει υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες, σε όλο τον πλανήτη. Δεν μπορούμε να ασχολούμεθα με τα πάντα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια χαρτοφυλάκια που θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγγύης Ανατολή είναι προτεραιότητα και επίση και το Αφγανιστάν είναι στι προτεραιότητε. Ειλικρινά, άμα δούμε 9 χρόνια μετά την αρχή του πολέμου στο Αφγανιστάν, το λιγότερο μπορούμε να πούμε είναι τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Ο πληθυσμό στο Αφγανιστάν πιστεύει ότι ουσιαστικά ο στρατό που είναι εκεί είναι ε, στρατό κατοχή. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη σήμερα, η ασφάλεια δεν είναι καλύτερη, ο αριθμό των πολιτών, των αμάχων που σκοτώνται σε αυτή τη σύγκρουση ε, αυξάνεται συνεχώ καθημερινά. Πληρώνουμε εκεί ε, για το ταμείο της Ανοικοδόμησης ε, στέλνουμε ευρωπαίου στρατιώτε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά στα πλαίσια οι μόνοι που αποφασίζουν για τη στρατηγική στο Αφγανιστάν είναι το ΝΑΤΟ. Το καταλαβαίνω, έχουν εντολή για να το κάνω αυτό. Αλλά εγώ σα ρωτώ το εξή. Ένα πράγμα τουλάχιστον. Τουλάχιστον να λάβετε μια πρωτοβουλία για πραγματικό προβληματισμό, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική όσον αφορά το θέμα του Αφγανιστάν. Ναι, αυτό σημαίνει ανάληψη κινδύνων. Πιθανότατα σημαίνει να μην περιμένουν και τι 7 κράτη-μέλη πάντα θα συμφωνούν επί των πάντων αλλά είναι πραγματικά ένα θέμα που απαιτεί να αναλάβουμε κάποιο κίνδυνο για να μπορέσουμε να, να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση τελικά που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Κούκαν, για 1,5 λεπτό, ο κύριος Κούκαν, πρόεδρος αντιπροσωπείας και εκείνο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πρόεδρε, Βαρονιά, στον ε, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε όλοι όταν τα πηγαίνετε καλά και ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά για τα Δυτικά Βαλκάνια, μία ερώτηση για την Βοσνία Ζεγοβίνη που δεν αναφέρθηκε. Ξέρω ότι η χώρα είναι δύσκολη και ξέρω ότι έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα αυτή. Έχετε νέες σκέψεις, νέες στρατηγικές για το τι θα πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη χώρα. Το ρωτώ αυτό γιατί θέλουμε να σας βοηθήσουμε να προάγετε να προωθήσετε νέες στρατηγικές, νέες τακτικές. Μία ερώτηση για το Ιράν, λίγο διαφορετική διατύπωση. Αναφέρατε μία διπλή προσέγγιση στο Ιράν. Χρειάζεται και το καρότο και το ε, μαστίγιο για την κατεύθυνση αυτή η, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καρότα έχουμε αρκετά. Μαστίγια όμως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα μισή λεπτό το επόμενο όνομα είναι Μύρσκι που έχω στο κατάλογο. Κύριος Μύρσκι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Λέδι Άστον. Σύμφωνα με ποιε αρχές κινείστε όταν διορίζετε τους πρεσβευτές για τη νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης διότι η Εστονία και η Λετωνία δεν εκπροσωπούνται αρκετά στη διπλωματική υπηρεσία της ευρωπαϊκής αυτής υπηρεσίας. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλή πρακτική. Τι θα κάνετε για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα. Μπραντνερ, η κυρία Μπραντνερ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε, Λεδιάστον. Δηλαδή, να θέσω ένα θέμα το οποίο αναφέρετε και προηγουμένως και καλωσορίζω τις προσπάθειές σας για την οικοδόμηση της ειρήνης, αλλά κοιτώντας τα γεγονότα, τα περιστατικά, ελπίζω να δω σύντομα να υπάρχει κάποιες νέες δομέ με κάποια διαμεσολάβηση σε υψηλό επίπεδο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάνουμε mainstreaming στην ε, οικοδόμηση της ειρήνης μέχρι ότι τελικά καταστεί ε, αναποτελεσματική. Γιατί χρειαζόμαστε κόσμο που να ξέρει τι κάνει. Κάτι άλλο που ήθελα να θέσω σε σχέση με τη Σομαλία. Είχαμε το εξής πρόβλημα. Έχουμε μια αποστολή στατιωτών ε, μάλλον ε, εκπαίδευση στρατιωτών και ξέρουμε ότι παράλληλα γίνεται εκπαίδευση και των, ε, της αντιπολίτευσης. Μια γερμανική εταιρεία εκπαιδεύει, ιδιωτική εταιρεία εκπαιδεύει τους, την αντιπολίτευση και η γερμανικό κράτος εκπαιδευτεί την εκπαίδευση της κυβέρνησης. Είναι περίεργο αυτό. Και βλέπουμε τι προβλήματα υπάρχουν στο Ιράν, στο Αφγανιστάν είναι γελίο το γεγονός ότι υπάρχουν απαστολές σε χώρες όπου υπάρχουν και δραστηριοποιούνται ιδιωτικέ εταιρείε προ την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό πραγματικά θα πρέπει να είναι μια πρωτοβουλία. Θα πρέπει να συζητηθεί επιτέλου το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. κυρία Ντεκάιζερ για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση του κυρίου Νταβίτ για τον Ταρέ Καζίζ. Μιλήσαμε εκτενώς στην ομάδα για τον πόλεμο στο Ιράκ. Μήπως ήρθα όμως ε, επιτέλους στιγμή να γυρίσουμε σελίδα. Δεν είμαι σίγουρη ότι η θανατική καταδίκη με απαχωνισμό του κυρίου Ταρέκαζής και άλλων δύο ατόμων δεν νομίζω ότι είναι ένας καλός τρόπος για να γυρίσουμε τη σελίδα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω το ρόλο που έπαιξε, δεν θα απονείμω εγώ δικαιοσύνη, αλλά πολύ είχαμε μεταβεί στο Ιράκ λίγο πριν τον πόλεμο, προσπαθώντας να προλάβουμε αυτό τον πόλεμο, να τον αποτρέψουμε. Είναι ένας άνθρωπος που είναι άνω των 70 πια, πέρασε από δύο εμφράγματα, καρδιακές προσβολές. Είναι πραγματικά ράκος αυτός ο άνθρωπος και αν αφήσουμε να εκτελεστεί θανατική ε, καταδίκη, από ανθρωπιστική άποψη είναι απαράδεκτο, δεν μιλάω για πολιτική. Θα ήθελα να σας δείσω να πραγματοποιήσετε διάβημα σχετικά. Είναι χριστιανός ο Ταρεκαζής. Είμαστε σε ένα πόλεμο Σουνιτών, Σιητών, Χριστιανών. Θα ήθελα λοιπόν να αποφύγουμε ένα νέο δράμα και οι εικόνες του απαχωνισμού του Σατάμ Χουσέιν που ήταν ένας άνθρωπος δικτάτορας και απεχθής άνθρωπος δεν κατέβνασαν τα πνεύματα στο Ιράκ ούτε ανακούφισαν τίποτα. Δεν νομίζω ότι μία ακόμη εκτέλεση θανατικής ποινής θα προσθέσει τίποτα. Λοιπόν, εσείς για τα συμπεράσματα, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, μέχρι τις 5 ώρα. Thank you uh, very much uh, again. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ντέιβιτ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σα για την ε, Ιορδανία. Ήταν καλή η συνεργασία με τον Υπουργό Εξωτερικών. Είμαστε νέοι συνεργάτες όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Να σα πω ευθύ ότι όσον αφορά τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, τον κύριο Αζής, είμαστε αντίθετοι προ τη θανατική ποινή. Όλη μου τη ζωή ήμουν κατά. Είναι ισχυρότατα τα συναισθήματά μου για αυτό το θέμα. Το γνωστοποίησαμε στην κυβέρνηση του Ιράκ θα πρέπει να ακολουθηθούν και άλλες διαδικασίες. Παρακολουθούμε προσεκτικότατα τις εξελίξεις. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας όσον αφορά τη σημασία. Ε, για τους πρεσβευτές για την υπηρεσία πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσία. Θα δείτε όταν θα αρχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία θα είναι σε επιχειρησιακή ε, φάση στι αντιπροσωπείε ε, θα βασιστούμε. Θέλουμε να είναι μια ευέλικτη, ευέλικτος μηχανισμός Βρυξέλλες που υποστηρίζει τις επιτόπου αντιπροσωπείες. Θα πρέπει να ενημερωθείτε όσον αφορά ε, ε, τα θέματα αυτά για να είστε σωστά ενήμερος. Κύριος Νόε, Δυτική Σαχάρα, Κνέου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα που δύο μέλη το έθεσαν το ζήτημα, διότι Γι' αυτό είναι και σημαντικέ αυτέ οι περιστάσει, γιατί και εγώ έχω τη δυνατότητα να δω τι έχετε υπόψη σα, τι έχετε στο μυαλό σα για τι περιοχέ του κόσμου. Κάναμε ένα γύρο του κόσμου, μεγαλύτερο από ό,τι θα νομίζαμε αρχικά. Προσπαθούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε, υποστηρίζουμε βέβαια τον Φερό, τον απεσταλμένο ότι ο ΟΗΕ για τον ρόλο του. Θα επισκεφθεί αυτό το μήνα, μάλλον από ό,τι γνωρίζω την περιοχή. Και ίσω θα ενημερωθούμε σαν επίσημε επαφέ μαζί του αλλά θέλω να εξετάσω το θέμα προσεκτικότατα, το δέχομαι το μήνυμά σας. Κύριε Πέτερλε, όλος ο χάρτης, δεν ξέρω αν καλύψαμε όλο τον χάρτη του κόσμου, αλλά σίγουρα είμαστε καθοδόν. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για τον Πιέρ Μορέλ, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός, ειδικό εκπρόσωπος, εργάζεται σκληρότατα και καθημερινά από το Κυρζικιστάν με ενημέρωνε όταν ξεκίνησαν οι ταραχέ. Συναντήθηκα με τον πρόεδρο όταν ήμουν στον ΟΗΕ στην ε, Γενική Συνέλευση. Συναντήθηκα μαζί τη, συζητήσαμε τα διάφορα θέματα που μα αφορούν. Προσπαθήσαμε να δώσουμε υποστήριξη, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή του κόσμου, έχετε δίκιο η ε, επίσκεψή μου στο Καζακστάν και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν μου έδειξαν ότι πρέπει να δούμε τι πόρους έχουμε για να είμαστε αποδοτικότεροι στην περιοχή. Γνωρίζω πολύ καλά τι κάνει ο Πιέρ και τον υποστηρίζω. Υποστηρίζω το έργο που επιτελεί εκ μέρους μας. κυρία Τεσάνες, το Αφγανιστάν, ανάληψη κινδύνων. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε κινδύνους που έχουμε συνειδητοποιήσει πολύ καλά και τους έχουμε αναλύσει. Δεν θέλω να κινηθώ κατά των 27 κρατών μελών, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω καμιά φορά να δίνω στα κράτη-μέλη ένα σχέδιο που θεωρώ ότι ίσως να είναι το ενδεδειγμένο. Αυτό που έχουμε στον κύριο Σουζάκης είναι ένας πολύ καλός ειδικό εκπρόσωπος που κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει μεγάλη φήμη. Πολλοί άλλοι εταίροι που ασχολούνται με το Αφγανιστάν μου το λένε σας είπα πως εκτιμώ τη σημασία που έχει η συνεργασία με τις γυναίκες του Αφγανιστάν και σημασία που έχει να μην φύγουμε από τις υποχρεώσεις που έχουμε λάβει. Παροχή, βοήθεια για τη δημόσια υγεία, υποστήριξη θεσμών, της παιδείας, επιβολής του κράτους δικαίου, όλα αυτά που είναι σημαντικά για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα στο Αφγανιστάν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να είμαστε εκεί. Ο κίνδυνος είναι να μείνουμε πολλοί για να δούμε να παγιώνονται αυτές οι εξελίξεις, πραγματικά ο κόσμος να μπορεί να ασχοληθεί με τη ζωή του και να προχωράει. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι όσον αφορά το πώς θα προσεγγίσουμε στο μέλλον το Αφγανιστάν. Ο κ. Κούκαν, Βοσνία Ερζεγοβίνη, σημαντικότατο θέμα, όπως είπατε. Το συζήτησα με την Υπουργό Εξωτερικών Κλίντον που είχε πάει πριν από 10 μέρες, όταν επέστρεψε και ήρθε στις Βρυξέλλες και θεωρούμε ότι είναι σημαντική στιγμή να προχωρήσουμε όσον αφορά τη στρατηγική μας με τη Βοσνία, να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε αυτή την κίνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 39% ανεργία τελευταία φορά που είδα τα στοιχεία, ολόκληρη γενιά νέων που χρειάζεται απασχόληση, ε, θέλει κάποιο μέλλον και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της η κυβέρνηση, να προσπαθεί να αναπτύξει μια ευρύτερη στρατηγική για το κάνουμε Έχουμε κάποιε ιδέε, ασχολούμαστε με το θέμα, Πεδιερευνήσω τι ιδέε περαιτέρω πριν τι ανακοινώσω, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σχετικά με το πώ θα προχωρήσουμε τι επόμενε εβδομάδε. Ιράν, μαστίγιο και καρότο, έχουμε αρκετά μαστίγια. Δεν έχω αμφιβολία στο μυαλό μου ότι το αποτέλεσμα των κυρώσεων είναι πραγματικό και ελπίζω, όπως είπα επανειλημμένα, ότι το Ιράν θα έρθει στο τραπέζι των συζητήσεων. Ο κ. Μόσκι, οι πρεσβευτέ, διορίζω του πιο έξυπνου, του καλύτερου. ξεκαθάρισα τη θέση μου όσο μπορούσα όσον αφορά τη γεωγραφική εκπροσώπηση, αλλά πρέπει να θυμηθείτε, έκανα μόνο ένα γύρο διορισμών πρεσβευτών βάσει μια διαδικασία που κληρονόμησα και δεν γνώριζα τι θα έκαναν τα κράτη-μέλη. Τώρα ξέρω τι κάνουν τα κράτη-μέλη και βλέπω τι ανάγκες υπάρχουν, πώς πρέπει να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά, πώς θα υπάρξει αυτό το γεωγραφικό εύρος, αυτό κάνουμε. Θα έχετε νέα όσον αφορά το θέμα αυτό, δεν μπορώ να τα κάνω με τη μία, σας το είπα. Χρειάζομαι χρόνο για να μπορέσω να αποδείξω ότι υπάρχει ευρεία κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να υπάρξει και κάλυψη του θέματος τη ισότητας των φύλων. Λίγη περισσότερη υπομονή σας ζητώ. Κυρία Μπράτνερ, ήξερα τι θα πείτε. Έχετε απόλυτα δίκιο εγώ υποστηρίζω και αυτά που είπα. Αυτό που κάνουμε είναι αποφυγή των συγκρούσεων και ε, δημιουργία ε, εμπιστοσύνη και ειρήνης. Αυτό είναι το λάβαρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πώς να αποφύγουμε τις συγκρούσεις, πώς υποστηρίζουμε τις διάφορες διαδικασίες της ανοικοδόμησης, πώ προσφέρουμε υπηρεσίε διαμεσολάβηση. Σερβία, κοσυφοπέδη, αν θέλετε. Προσπαθούμε να το κάνουμε στην πράξη αυτό. Αυτό προσπαθώ να κάνω και θέλω να είμαι σίγουροι ότι έχω του ανθρώπου στη διάθεσή μα. Αλλά αυτό θέλουμε σίγουρα ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό το λόγο προβάλλω αντιρρήσει Να, δεν θέλω να δίνω τίτλους σε διάφορα κομμάτια του οργανισμού, αλλά το σύνολο. Ξανά θα έχω νεότερα αργότερα. Δεν ξέρω για το θέμα των ιδιωτικών εταιριών ε, ασφαλείας. Είναι πολύ σημαντικό σίγουρα. Το συζητήσαμε και αυτό με τους επικεφαλείς των επιτελείων πρέπει να γίνει σωστή προσέγγιση όσον αφορά τις επιτόπιες δομές. Ευχαριστώ που το θέσατε, το ζήτημα είναι σημαντικό. Και κυρία Ντεκάιζερ, νομίζω ότι απάντησα το ερώτημά σας σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στο Ιράκ και το θέμα της θανατικής ε, καταδίκης, της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ, είπα τη εκπρόσωπε, όχι μόνο για το περιεχόμενο, αλλά και για τη μέθοδο που ακολουθήσατε, υπήρξατε, ακριβέστατη συνοπτικότατη και ευγενέστατη εκφράσατε κάποιες σκέψεις όπως και εμείς, κάποιους προσανατολισμούς, κάποιες χρήσιμες ειδήσει μας δώσατε, έχοντας ακούσει τους συναδέλφους και νομίζω ότι αυτά υπήρξαν χρήσιμα και χρήσιμα και για την ευαίσθητη δουλειά σας. Ήταν χρήσιμα και για μας, ανανεώνουμε την πρόσκλησή μας για να επιστρέψετε εδώ σύντομα να μας βρείτε όταν θα υπάρξουν και σίγουρα άλλες εξελίξεις σημαντικές προσχολιασμών και προτάσεις να παραλάβετε και να δώσετε. Σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά και στο επανειδήν σύντομα. Σε πέντε λεπτά θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Παρακαλώ να παραμείνετε στις θέσεις σας, να καθίσετε στις θέσεις σας μάλλον. Λοιπόν, έχουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη τη δημόσια κρόαση όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς στα Δυτικά Βαλκάνια. Η επιλογή έγινε για τη διεξαγωγή αυτής τη ακροάσεως από τα ερωτήματα που θέσαμε, δηλαδή τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την κρίζωση της ε, ε, διαφθοράς από την άμεση γειτονιά μας. Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Θελήσαμε να δώσουμε μια προοπτική προς ευρωπαϊκή ένταξη σε αυτή την περιοχή. Το κράτος δικαίου είναι βασική αρχή που πιστεύουμε είναι ουσιαστική αξία και επαναλάβαμε ότι η δημοκρατική οικονομική ανάπτυξη ε, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ αυτών κυρίως σημαντικός όρος είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Πολλές προσπάθειες ήδη έχουν καταβληθεί για να εφαρμοστούν πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς. Κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πιο συγκεκριμένα και σημειώσαμε και τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς τις επιτυχίες που επετέφθησαν. Όλα αυτά επετέφθησαν όταν η συνεργασία ήταν πολιτομιακή ούτως πίν. Με της κυβερνήσεως, του επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, όλοι μαζί, συντονισμένοι, συνεργαζόμενοι, καθορισμός προτύπων διαδικασιών και υποστήριξη για την επίτευξη των κοινών σκοπών. Η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν εξαντλείται με μια χειρονομία και σε μια κίνηση. Χρειάζεται μια συνεχής ε, κινητοποίηση, συνεχής προσπάθεια για να μπορέσει κανείς να πετύχει τα ευθεία αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε σήμερα να συμβάλλουμε στη διαδικασία, στην προσπάθεια, σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται, μέσω ενός βήματος συζητήσεων, και καλέσαμε για αυτό το φόρουμ εμπειρογνώμονες σημαντικούς που γνωρίζουν καλά την περιοχή για μια ανταλλαγή απόψεων για να συζητήσουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές της περιοχής για κάθε χώρα μάλλον και τι γίνεται για την καταπολέμηση της διαφθοράς. για να γνωρίσουμε πώς δημιουργείται το φαινόμενο, τα χαρακτηριστικά του και πώς να καταπολεμηθεί είναι προϋποθέσεις αυτές που ανέφερα για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσει η κυρία Τεζέβα, πρόεδρος του Zero Corruption Macedonia, όσον αφορά τις προοπτικές της περιοχής και των χωρών όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μετά η κυρία Κάλοβιτς του Μαντς Μοντενέγκρο, για να συζητήσουμε το πώς μπορεί να... τι γίνεται με την καταβολή της διαφθοράς στο, Μαυροβούνιο. Και τρίτον, ο κύριος Ντερβίση που θα περιγράψει την κατάσταση στην Αλβανία. Θα ακολουθήσουμε αυτή τη σειρά. Θα σας παρακαλούσα, αν μπορείτε, να τηρήσετε ένα δεκάλεπτο ο καθένας όσον αφορά τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, η, κυρία, η καθηγήτρια Ταζέβα. Η κυρία Ταζέβα. Thank you, Mr. Albertini. Σας ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη που νιώθω για την πρόσκληση σε αυτή την επιφανή ομίγυρη και ευελπιστώ ότι θα μπορέσω να συμβάλλω κι εγώ μαζί με τους συναδέλφους στην εμβάθυνση του προβλήματος της πάταξης της διαφθοράς στα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω ότι στην αρχή δεν θα έχω PowerPoint, με, αφού κατέπτυσα τους πίνακες όμως είπα ότι μιλάνε από μόνοι τους. Καλύτερα λοιπόν να τους προβάλλουμε οθόνες για να είναι πιο ορατή η κατάσταση της διαφθοράς της χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και για όσους παρακολουθούν την ακρόαση. Θα κάνω καταρχήν κάποιες αναφορές σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του δίκτυου διαφθοράς που δημοσιεύθηκαν χθε, όπως θα ξέρετε και έγινε εξή ταξινόμηση. Η Δημοκρατία της Μακεδονίας μαζί με την Κροατία βρέθηκαν στην 62η θέση το Μαυροβούνιο στην 69η, η Σερβία στην 78η, η Αλβανία, η Αλβανία στην 87η, η Βοσνία στην 91η και το Κωσυφοπαίδιο στην 110η θέση. Για πρώτη φορά συμπεριληφθήκε στο κατάλογο και σχεδόν όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έδειξαν βελτίωση και πρόοδος ό,τι αφορά τη θέση τους ε, στη... στον κατάλογο ε, της διαφθοράς αλλά είναι σημαντικά ε, τα μόρια της διαφθοράς και όχι θέση. Για παράδειγμα, η Μακεδονία ανέβηκε από την 72η στην 69η θέση. Δεν ήταν σημαντική αυτή η διαφορά στις θέσεις, αλλά η διαφορά στη, στα index points ήταν μόνο 0,3. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η λήψη υπόψη των δικτών, όχι η θέση στον πίνακα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τη θέση των ευρωπαϊκών χωρών σε σύγκριση με την Τουρκία, που επίσης είναι υποψήφια χώρα σε αυτό τον κατάλογο. Βλέπουμε ότι ακόμη και μερικές ευρωπαϊκές χώρες μέλη βρίσκονται πολύ χαμηλά στον κατάλογο για, για το δίκτυ διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτού του πίνακα από το 2007, 2008, 2009 και 2010 για τα Δυτικά Βαλκάνια, είναι χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τις διαφορές και τις βελτιώσεις. Μία θεαματική βελτίωση φαίνεται συγκρίνει με τα διάφορα χρόνια. Σκούρο μπλε είναι το 2007 και το 2010 είναι ένα ανοιχτό γαλάζιο. Θα διαπιστώσετε ότι όλες οι χώρες στην περιοχή έδειξαν κάποια πρόοδο. Βλέπετε ότι ανήλθαν στον κατάλογο ταξινόμηση ό,τι αφορά το δίκτυ εντοπισμού διαφθοράς. Η διεθνής διαφάνεια προβαίνει στην κατάρτιση αυτού του πίνακα και διαπιστώνει ότι υπάρχει βελτίωση στις διάφορες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η διεθνής διαφάνεια χρησιμοποιεί και ένα άλλο μέσο για να αποτιμήσει τη διαφάνεια. Πρόκειται για το βαρόμετρο της συνολικής διαφθοράς που στηρίζεται σε εμπειρικά στοιχεία, σε αντίθεση με τους δείκτες, και στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία της ε, δημολογικής απογραφής και στις ερωτήσεις υπάρχει ερώτηση πότε σας ζητήθηκε φακελάκι πότε σας ζητήθηκε προμήθεια ή πότε χρειάστηκε να δωροδοκίσετε κάποιον για να εξυπηρετηθείτε τα αποτελέσματα από αυτή την δημοσκόπηση διαφέρουν από τα αποτελέσματα του δίκτυ διαφθοράς, αντίληψης της διαφθοράς. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε το δίκτυ διαφθοράς και στην άλλη περίπτωση έχουμε την προσωπική εμπειρία των ανθρώπων. Είναι και θέμα βέβαια εμπιστοσύνης του λαού στην κυβέρνηση του κάθε φορά κατά πόσο ο λαός πιστεύει ότι η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική στην πάταξη της διαφθοράς. Βλέπουμε ότι στη Μακεδονία οι πολίτες έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή τους και πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους θα πάει καλά στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις εμπιστοσύνης τις έχει η Βοσνία Ζεγοβίνη. Βλέπετε και τις επιδόσεις ε, της Κροατίας και της Σερβίας, που επίσης είναι χαμηλά προς την εμπιστοσύνη του λαού στην άρχουσα τάξη. Τώρα, αν εξετάσουμε τις διαφορετικές κατηγορίες αξιωματούχων, των πολιτικών κομμάτων, ε, των επιχειρήσεων, διδικοτικού κλάδου, δημοσίων υπαλλήλων και δικαστών και στην ερώτηση σε ποιο βαθμό μια κατηγορία συνέβαλε στη διαφθορά στις αντίστοιχες χώρες, βλέπετε ότι ισχύει σχεδόν το ίδιο σχήμα στον πίνακα. Η βασική κατηγορία που πειράζεται από τη διαφθορά είναι τα πολιτικά κόμματα και οι κάτοικοι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης πιστεύουν ότι η πολιτική τους, ότι τα πολιτικά κόμματα είναι άκρως διαφθαρμένα. Το ίδιο ισχύει και για τη Σερβία. Στη Μακεδονία, την Κροατία, το Κωσυφοπαίδιο και το χαμηλότερο σκορ το βλέπουμε στην Τουρκία. Το ίδιο pattern έχουμε και εδώ και για τις επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Στη Βοσνία πιστεύει ο κόσμος ότι οι επιχειρήσεις είναι διεφθαρμένες. Το ίδιο ισχύει και για την Κροατία. Σήμερα ακολουθεί η Σερβία, η Μακεδονία και το Κωσυφοπαίδιο. Δημόσια διοίκηση, δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν χαίρουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη ούτε στη Βοσνία ούτε στην Κροατία και μετά Κροατία, Σερβία για το δικαστικό κλάδο. Ίδιο σχήμα και εδώ. Ο κόσμος έχει αντιμετωπίσει προβλήματα διαφθοράς ακόμη και στο δικαστικό κλάδο στην πατρίδα τους. Το πρόβλημα βέβαια της διαφθοράς ε, μόνο στην Τουρκία δεν θεωρείται ως μείζον στο δικαστικό κλάδο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Αν ε, ρωτήσαμε τον κόσμο αν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για να αγοράσουν από μία ε, επιχείρηση που δεν έχει ιστορικό διαφθοράς. Βλέπετε που ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πληρώσει έστω και ακριβότερα σε μια καθαρή επιχείρηση. Αυτά ως προς το βαρόμετρο της συνολικής διαφθοράς που μας δίνει μία εντύπωση για το ποια είναι η γνώμη του λαού για, το φαινόμενο της διαφθοράς στη χώρα. Και έχουμε και μία συγκρίση μεταξύ των χωρών της περιοχής. Έγιναν και άλλες μελέτες όμως για την περιοχή που αφορούν το πρόβλημα του εγκλήματος και της διαφθοράς στα Δυτικά Βαλκάνια. Μία από τις μελέτες είναι η Βαλκανική μελέτη του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2008 με βάση τη μελέτη αυτή, ενώ το επίπεδο ε, συμβατικού εγκλήματος στα κράτη-μέλη αυτά φαίνεται, στα κράτη αυτά φαίνεται ότι μειώνεται, μόνο μία εγκληματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα προβληματική στα Βαλκάνια, είναι η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα. Αυτό ε, είναι το συμπέρασμα της βαλκανικής μελέτης ε, των Ηνωμένων Εθνών. Βέβαια είναι δύσκολο να καταμετρηθεί η έκταση αυτού του φαινομένου, αλλά έχουμε την περίπτωση των δωροδοκιών, φακελάκια και απάτη κατά το καταναλωτή. και έχουμε τα περισσότερα θύματα. Υπάρχει και πρόβλημα με τις καταγγελίες Το πρόβλημα δυστυχώ δεν μειώνεται. Τι κάνουν όμω οι χώρε για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Αρκετά, πολλά θα έλεγα. Και χάρη στη διεθνή συνεργασία, οι χώρε τη περιοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης, γιατί όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι μέλη και του Γκρέκο και του Συμβουλίου της Ευρώπη. και συμμετέχουν σε πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Και μάλιστα με την ε, έναρξη της διαδικασίας ε, σύνδεσης και ένταξης για πολλές χώρες των Δυτικών Βαλκανίων γίνονται σημαντικές προσπάθειες για εναρμόνιση της νομοθεσίας τους ε, στο θέμα της πάταξης της διαφθοράς. Βλέπουμε όμως στην έκθεση πρόοδου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2007 αλλά και την έκθεση του 2009 Βλέπουμε ότι οι Βρυξέλλες, ε, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει πολλές επικρίσεις ό,τι αφορά την ε, χαμηλή πρόοδο, ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς, ιδιαίτερα στο δικαστικό κλάδο. Σε ό,τι αφορά τις ε, εσωτερικές δραστηριότητες, είδαμε κάποια αναρμόνιση της νομοθεσίας σχεδόν σε όλες τις χώρες που έχουν προσυπογράψει και κυρώσει την συνθήκη UNCAC. Βέβαια υπάρχουν διαφορετικές εσωτερικές νομοθεσίες ε, και αντίστοιχες ε, εφαρμόζουν και τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουν αναπτύξει και ε, στρατηγικές καταπολέμησης της διαφθοράς και πολλές χώρες αναθεωρούν τα προηγούμενα προγράμματα δράσης και τα ενημερώνουν προκειμένου να γίνουν πιο δραστήρια και μάλιστα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σε όλες ε, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχουν και φορείς, ε, οι οργανώσεις, ε, ειδικά σώματα κατά της διαφθοράς. Υπάρχουν σε όλες τις χώρες ειδικοί οργανισμοί καταπολέμησης της διαφθοράς και σε ορισμένες χώρες, τη Σερβία, τη Μακεδονία, το Κωσυφοπαίδιο, αυτές, αυτοί οι οργανισμοί έχουν ιδρυθεί ως ανεξάρτητα ιδρύματα με ξεχωριστή νομοθεσία και μάλιστα στο Μαυροβούνιο είναι ένα προεδρικό διάταγμα που θέσπισε αυτή την, ε, αυτή την ε, υπηρεσία, ενώ στην Κροατία υπάρχει το ΟΥΣΚΟΚ που είναι τμήμα ε, του Γενικού Εισαγγελέως της ε, Κρατικής Εισαγγελικής Αρχής. Το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά τα σώματα πάταξη διαφθοράς ή τους οργανισμούς είναι ότι έχουν μικρό, λίγο προσωπικό, δεν έχουν επαρκή σπόρους, δεν έχουν επαρκή τρόπο συλλογή στοιχείων και κατάλληλη συνεργασία με τις χώρες, με το Κοινοβούλιο. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που επισημαίνει η έκθεση Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η έλλειψη εφαρμογής η ελλειπή εφαρμογή τη ε, νομοθεσία. Η νομοθεσία υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Αλλά και η κοινωνία των πολιτών δεν έχει ούτε πόρου ούτε και δύναμη για να ασκήσει τον έλεγχο και να υποστηρίξει τι δραστηριότητε πάταξη τη διαφθοράς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο διευκόλυσης των δραστηριοτήτων καταπολέμησης διαφθορά και βιωσιμότητα του κράτου δικαίου στι χώρε αυτέ. Ένα από του τρόπου ίσω θα ήταν κάποιε κοινέ δραστηριότητε για την εφαρμογή της συνθήκης UNCAC και της Ευρωπαϊκής Συνταξιακής Διαδικασίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τάσεβα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και τηρήσατε και το χρόνο σας. Κυρία Τσάλοβιτς, έχετε το λόγο. Σας θέλω, παρακαλώ, μην ξεπεράσετε και εσείς το δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Μπάνια Τσάλαβιτς ονομάζομαι, Για το Μαυροβούνιο έρχομαι και εργάζομαι κατά των ε, συμφερόντων της κυβέρνησής μου και των πολιτών μου, όπως αναφέρει η κυβέρνησή μου, αλλά και πάλι οι πολίτες αναφέρουν ότι εμπιστεύονται πιο πολύ εμένα παρά οποιονδήποτε πολιτικό στη χώρα μου. Το Μαυροβούνιο μοιάζει πολύ, αλλά παρόλα αυτά διαφέρει από τις άλλες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι η μοναδική χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, η μοναδική χώρα μετά τον κομμουνισμό που δεν άλλαξε την κυβέρνησή της. Έχουμε ακριβώς τις ίδιες δομές κυβερνητικές εδώ και δύο δεκαετίες. Ακόμα και αν ήταν η καλύτερη κυβέρνηση που υπήρξε ποτέ, ακόμα και αν η πολιτική ήταν η πιο ειλικρινής και τίμη, ακόμα και αν είχαμε ε, αντιπολίτευση ισχυρή και ισχυρή πολιτεία των ε, ε, κοινωνία των πολιτών θα υπήρχε κάποια διαφθορά μετά από 20 χρόνια. Ιδιαίτερα επειδή περάσαμε και από πόλεμο, περάσαμε κυρώσεις κατά την περίοδο εκείνη. Ε, έλαβαν χώρα διάφορες, ε, για παράδειγμα, λαθρεμπόριο τσιγάρων, διάφορα πράγματα τα οποία θα τα θεωρούσαμε ως ε, εγκλήματα. Δεν κόψαμε λοιπόν τις σχέσεις μεταξύ της εκτελεστικής μας εξουσίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν υπάρχει ούτε ένα αφεστό σε ολόκληρο τον κόσμο που να υπάρχουν τέτοιες ελίτ, οι οποίες πρόθυμα και ειλικρινά να ξεκίνησαν να καταπολεμήσουν τα κυκλώματα λαθρεμπορία στα οποία η ίδια, τα, ίδια τα, κυκλο, τα ίδια συστήματα είχαν συστήσει. Σύμφωνα με την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Μαυροβούνιο παραμένει βασικός κρίκος της αλυσίδας λαθρεμπορίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Ωστόσο, το Μαυροβούνιο είναι και ασυνήθιστο για έναν άλλο λόγο που ανέφερε και η συνάδελφος Απαντήσαμε σε κάποιες ερωτήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φάνηκε ότι θεωρούμε ότι έχει αυξηθεί η διαφθορά. Ωστόσο αυτό δεν ε, ανταποκρίνεται με τις μεταρρυθμίσεις, γιατί ε, θεωρεί ο κόσμος ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη διαφθορά φέτος από ότι στα προηγούμενα χρόνια. και η ελευθερία των μέσων είναι αμφισβητήσιμη. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι το Μαυροβούνιο είναι η μοναδική χώρα η οποία κρατάει την εφαρμογή του κοινωτικού κεκτημένου κρυφή και από το Κοινοβούλιο και από τους πολίτες τους ίδιους. Καταφέραμε να μάθουμε τέτοια στοιχεία, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ασκήθηκαν πιέσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ρώτησε η Κομισιόν πόσα χρήματα λάβαμε από την ιδιωτικοποίηση και μας είπαν τόσο από τη μία εταιρεία ε, τόσα από την άλλη εταιρεία, αλλά δεν μας είπαν πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά και το ρώτησε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξαναρώτησε η Επιτροπή λοιπόν, αλλά δεν πήρε απάντηση. Τρεις φορές ρώτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά και τρεις φορές δεν έλαβε απάντηση. Γιατί, γιατί η κυβέρνηση δεν ήθελε να συμμετάσχει περισσότερος κόσμος στην διαδικασία της ένταξης στην Ένωση, γιατί θέλουν να αποφύγουν τέτοιες ερωτήσεις και ουσιαστικά προσπαθούν να ξεγελάσουν τη διεθνή κοινότητα και προσπαθούν να υποκριθούν ότι δεν είναι τόσο προβληματική η περίπτωση του Μαυροβουνίου όσο στη Σερβία, του Κωσυφοποδίου και το καθεξής. Γιατί όμως ήταν έχει αλλάξει η κυβέρνηση στο Μαυροβούνιο. Άρα θεωρεί, ίσως ε, θεωρούν η κυβέρνηση ότι θα θεωρήσουν οι Βρυξέλλες ότι είναι σταθερή η κυβέρνηση και ότι είναι καλή η κυβέρνηση επειδή είναι σταθερή. Μία άλλη πρακτική ε, στο Μαυροβούνιο είναι να κάνουμε κατάχρηση της κοινωτικής ε, ε, διαδικασίας. Οποτεδήποτε συμβαίνει κάτι κακό, δεν είναι προνομιακή συμπεριφορά, για παράδειγμα προς κάποιους επενδυτές, η δικαιολογία που χρησιμοποιείται είναι ότι α, το κάνουμε για να συνάδουμε με το κοινοτικό κεκτημένο. Και μια, ένα χρόνο αργότερα λαμβάνουμε την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλες αυτές οι διατάξεις δεν συνάδουν με το κοινωτικό κεκτημένο. Κάτι άλλο, το οποίο είναι επίσης ασυνήθιστο για το Μαυροβούνιο και θεωρώ ότι πολλοί πολιτικοί από εσά, ε, αν γνωρίσετε μέλη της πολιτικής μας ελίτ, είναι η πιο φτωχή πολιτική που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου να υπάρχουν. Στο όριο της ένδυας ε, ζουν. Α, βέβαια, το τρόπο ζωής τους δεν συνάδει με αυτά που επίσημα δηλώνουν, αλλά σύμφωνα με τις επίσημα στοιχεία, το Μαυροβούνιο είναι η μοναδική χώρα που έχει το τόσο ψηλό, τόσο μεγάλο χάσμα ένδυας. Και αυτά συνέβησαν μετά την ιδιωτικοποίηση, γιατί η ιδιωτικοποίηση δεν ε, απέφερε τα, τα ε, αναμενόμενα ε, κέρδη, δεν έφερε επενδύσεις, δεν έφερε εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε όλο και πιο πολλές κοινωνικές αναταραχές, διαμαρτυρίες, απεργίες, οι οποίες απειλούν τον κόσμο, ο οποίος τι θέλει, θέλει νέε επενδύσεις, θέλει ε, κατά δεύτερον να γίνονται σεβαστά τα εργασιακά δικαιώματα. Δυστυχώς, από, επειδή η κυβέρνηση δεν ακούει τις διαμαρτυρίες αυτές, όλο και πιο πολλοί κόσμος ε, ε, χάνει σκεύον τη ζωή του, τέλος πάντων απειλείται η ζωή του με απεργίες πείνας και ούτω καθεξής. Οι πιο πολλοί επενδυτές που ήρθαν στη χώρα έρχονται από μία χώρα, τη Ρωσία. Και γι' αυτό το Μαυροβούνιο αποκαλείται συχνά η Μόσχα η παράκτια. Χτες, ο Υπουργός Εξωτερικών μας, από τον ε, Ρώσο ομολογό του, έλαβε ένα μήνυμα για την συμβολή του για την διεθνή συνεργασία και να σας πω ότι ο υπουργό μας έκανε πολύ καλή δουλειά γιατί η πλειοψηφία των ε, Ρώσων επιχειρηματιών κινούν περισσότερο από το ίμιση της οικονομίας μας. Και καταστρέφουν το περιβάλλον σε μια χώρα όπου υπάρχει σύνταγμα και αναφέρεται ως οικολογική χώρα. Δυστυχώς όλοι οι θεσμοί ουσιαστικά αγνοούν την ύπαρξη των παράνομων αυτών δομών και αγνοούν τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος στις οικοδομές. Έχουμε μόνο... Δεν υπάρχει καμία περίπτωση δικαστικής ε, εκδίκασης ε, περιπτώσεων ξεπλήματος χρήματος. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στο μαύρο βόνιο αλλά για να ικανοποιήσουμε εσάς και την Ουάσιγκτον η κυβέρνηση παίζει με τα στατιστικά στοιχεία για τη διαφθορά, γιατί αναφέρεται για παράδειγμα ότι δεν υπάρχει στην αστυνομία Αναφέρεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στην διαφθορά σε υψηλό ή σε χαμηλό επίπεδο, για παράδειγμα, στην αστυνομία. Εμείς ποτέ δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Ο καθημερινός ε, κόσμος που δεν πληρώνει φόρους, η αστυνομία, αυτούς ε, μάλλον ε, κυνηγάει η αστυνομία για να βγάλει τα στατιστικά στοιχεία που χρειάζεται. Επίσης να σας πω ότι στις άλλες ε, χώρες κάνουν μέρος της δικής μας δουλειάς. Για παράδειγμα, η Κροατία, η Σερβία εξετάζει δομές παράνομης εμπορίας κοκαίνης μέσω του Μαυροβανιού και μιλάω για πάνω από 3.000 κιλά κοκαίνης. Η Μακεδονία επίσης κάνει δική μας δουλειά και πάλι εκδιώκουν ε, παράνομους λαθρέμπορους, λαθρέμπορους μάλλον κοκαίνης. Αλλά ακόμα και αν αποδεικνύουμε ότι υπάρχει κόσμος στη δημόσια διοίκηση που σχετά στενά σχετίζεται με διαφθορά και πάλι δεν κάνουν τίποτα. Κάποιος ε, δημοσίευσε ένα βίντεο γάμου ενός σημαντικού επιχειρηματία από ένα άτομο το οποίο κάνει λαφρεμπόριο ερωίνης και το βίντεο αυτό αποδεικνύει ότι όχι μόνο γιορτάζουν μαζί τέτοιοι εγκληματίε, αλλά και ότι οι υψηλοί αξιωματούχοι της μυστικής υπηρεσίας γιορτάζουν μαζί τους, ε, ε κάνουν πλάκα, τους φιλάνε. Σε ποια άλλη χώρα δεν θα γινόταν έρευνα για το τι κάνει ο αξιωματούχος αυτός της μυστικών υπηρεσιών με τους εγκληματίε και έρχονται και μας ανακρίνουν εμά. Αν ξέρουμε ποιος έβγαλε στο ίντερνετ το βίντεο, ανακρίνουν τους δημοσιογράφους για το ότι μιλάνε. Έτσι καταπολεμούν τη διαφθορά, καταπολεμούν εκείνους που θέτουν ερωτήσεις για το οργανωμένο έγκλημα και για να κλείσω να σας πω ότι πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο δεν έχει εμπειρία σε ούτε έναν τομέα στη διαφθορά. Έχουμε μεγάλες ομάδες, μικρές ομάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τη δημόσια διοίκηση για να την χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Αν το Μαυροβούνιο δεν κάνει καμία πρόοδο προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, αν μας πείτε ότι είστε η Κολομβία των ε, Βαλκανίων και δεν σας θέλουμε, μόνο οι κακοί τελικά θα ωφεληθούν από, αυτό. Μόνο οι κακοί θα ωφεληθούν από οποιαδήποτε αναβολή της ε, κοινωτικής, της ε, ενταξιακής διαπραγμάτευσης. Σας ευχαριστώ κύριε Κάλοβιτς. Ο κύριος Τερβίση έχει το λόγο για να μιλήσει για την κατάσταση στην Αλβανία για 10 λεπτά ενδεχομένως. Θα σας μιλήσω για 10 λεπτά. Λούτφιντερ Δερβίση ονομάζομαι και τα τελευταία 20 χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Εργαζόμουν ως δημοσιογράφος. Όταν η γυναίκα μου όμως είπε στον γιο μου ότι πρέπει να διαβάσεις το σχολείο γιατί αλλιώς θα καταλήξεις σαν πατέρα μου, στον πατέρα σου, άλλαξα επάγγελμα. Η Αλβανία σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, την διαφάνεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς, από το 2001 έχουμε, λαμβάνουμε εκθέσεις πρόοδου, όπου δύο προτάσεις παραμένουν σχεδόν απαράλλαχτες κάθε χρόνο. Η διαφθορά παραμένει σημαντικό πρόβλημα για την Αλβανία και στην Αλβανία δεν υπάρχει πρόβλημα με την ε, εκδίκαση, με τη θεωρία, αλλά με την εφαρμογή των, ε, της νομοθεσίας για τη διαφθορά. Υπάρχει έντονη... Ε, το κοινό πιστεύει ότι υπάρχει έντονη διαφθορά και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα που ακόμα και το δικαστικό σώμα πληρώνει το τίμημα της πολιτικής διαφθοράς. Οι πολιτικοί ανησυχούν για την αμοιμότητα και ζητούν την, επιζητούν την ε, υποστήριξη του κοινού και ανησυχούν και για την διεθνή κοινότητα, αλλά και το κοινό το απασχολούν οι διεθνείς οργανώσεις. Μία παρτηρήση για τις εκτάσεις πρόοδου. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με προτάσεις όπως ε, έχει γίνει πρόοδος αλλά χρειάζεται παραπάνω πρόοδος. Γιατί κάποιοι πολιτικοί διαβάζουν μόνο το πρώτο τμήμα, η πολιτική της κυβέρνησης. Ενώ οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης διαβάζουν το δεύτερο τμήμα της πρότασης. Μας απασχολεί η διαδικασία ένταξης στην Ένωση. Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, οι Αλβανοί εμπιστεύονται πιο πολύ τις δημόσιες, τις ε, παγκόσμιες ε, οργανώσεις, τον ΝΑΤΟ, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά τον Πρόεδρο της στρατιωτικές οργανώσεις, το δικαστικό σύστημα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τέλος, τέλος, τον πάτο της λίστας είναι τα πολιτικά κόμματα. Για να το σκεφτούμε αυτό. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ της αντίληψης που επικρατεί στον κόσμο για τη διαφθορά και της εμπιστοσύνη. 89% των Αλβανών θα έλεγε ναι στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μεγάλες οι προσδοκίες για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για θέματα ταξιδίου και για τις θεωρήσεις. 87% των Αλβανών λένε ότι αποδέχονται ότι θα ενισχυθεί ε, το κράτο δικαίου. 85% θεωρεί ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα και 61% περιμένει πιο πολλές ε, δραστηριότητες οικονομικές. Και 75, 77% θεωρεί ότι θα υπάρχει λιγότερη διαφθορά. Μετά το 97 η διαφθορά έγινε πολύ αγαπητό θέμα στην ε, Αλβανία, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα στην κορυφή της ατζέντα των προτεραιοτήτων. Η λειτουργία των δομών, η σταθερότητα και τελευταία αναφέρεται παντά η διαφθορά. Κοιτώντα τι έγινε τα τελευταία δέκα χρόνια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Καταρχά έγινε μια προσπάθεια για καλή διακυβέρνηση και αυτό το βλέπουμε και από τα πρώτα project που εφαρμόστηκαν 2000-2005 και που επικεντρώθηκαν στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στο κράτος δικαίου και στους νέους ε, νόμους και όχι τόσο για μέτρα κατά της διαφθοράς. Άλλη μια σημαντική συμβολή είναι ένα κοινό project της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρόσφατες επιτυχίες τώρα. Να σας πω μία από τις πιο σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις της δημόσιας δίκαιης είναι κάποιες ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Νομίζω ότι η Αλβανία είναι μια μοναδική χώρα με 100% σχεδόν ηλεκτρονική, ηλεκτρονικό σύστημα ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης ε, υπάρχουν ε, ειδικέ υπηρεσίε πολέμηση και πάταξη τη διαφθορά. Αυτό όμω δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική θέληση, μάλλον την έλλειψη πολιτική θέληση. Αναλύοντα την πολιτική διαφθορά, διαγράφονται κάποια αρνητικά κάποιες αρνητικές εξελίξεις. Καταρχάς, δεν έχουν βρεθεί λύσεις για την πλειονότητα των ε, περιπτώσεων διαφθοράς και των σχετικών κατηγοριών. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τις σχετικές διαδικασίες. Κατά δεύτερον, πολλές σχετικές κατηγορίες γίνονται μετά από εκλογές και σε πολλές περιπτώσεις ε, αναφέρεται ότι οι κατηγορίες αυτές ήταν ψέματα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αφιλία, ασυλία. Τα κόμματα υφίστανται χωρίς τους απαραίτητους κανόνες διαφάνειας για τα οικονομικά τους και μια προβληματική κατάσταση είναι επίσης ο διορισμός των δημοσίων υπαλλήλων. Η διαρκής αλλαγή των δημοσίων υπαλλήλων ανάλογα με την κυβέρνηση και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώ. Το δικαστικό σώμα εξακολουθεί να πλήττεται από διάφορα προβλήματα. Καταρχάς, ότι υπάρχει ακόμα το παλιό κομμουνιστικό σύστημα και σήμερα έχουμε διαφορετικό σύστημα, αλλά ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του δικαστικού συστήματος προκύπτει από το παλαιό σύστημα. Κατά δεύτερον, το δικαστικό σύστημα, η δικαστική τάξη έχει στενές σχέσεις με την πολιτική τάξη. Δεν υπάρχουν επαρκείς διοικητικές ε, ποινές για τους δικαστές. Χάρη στις ιδιαιτερότητες του δικαστικού συστήματος, ουσιαστικά είναι συμβολικής ε, φύσεως οι δυνατότητες που υπάρχουν κατά των δικαστών. Κατά τρίτον, δεν υπάρχει σύστημα για να διασφαλιστούν οι επαγγελματικές ικανότητες των δικαστών. είναι ουσιαστικά εγγυημένη η διαφθορά των δικαστών, καθώ δεν έχουν και επαρκή χρηματικο... αμοιβέ. Δεν έχουν επαρκή αμοιβέ. Όλοι αυτοί οι παράγοντε έχουν δημιουργήσει ένα δικαστικό σώμα το οποίο δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο στην καταπολέμηση και πάταξη τη διαφθορά για το ρόλο τώρα των μέσων μαζική ενημέρωση σε ό,τι αφορά την διαφθορά. Στην Αλβανία υπάρχουν περίπου 30 εφημερίδε, 4 κανάλια, 4 ψηφιακές πλατφόρμες και παραπάνω από 12 ψηφιακά κανάλια. Και όλα αυτά φυσικά συμβάλλουν στη δημόσια συζήτηση. Δεν χάνουμε σχεδόν κανένα ανακοινωθέν τύπου. Θεωρούμε ότι είναι θεματοφύλακα ε, τα μέσα αλλά να σα θυμίσω ότι ποτέ δεν γαυγίζουν οι σκύλοι όταν περνάει μέλο τη οικογένεια του από δίπλα. Έχουμε μέσα μαζική ενημέρωση ε, που τάσσονται με την κυβέρνηση και άλλα που τάσσονται με την αντιπολίτευση. Οι μάνοι κατηγορούν του δε. Και οι κατηγορίες για τη διαφθορά φεύγουν κατευθείαν από τους πολιτικούς ηγέτες και μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να έχουν καν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών τώρα. Κοιτώντα τι γίνεται γενικά στην κοινωνία των πολιτών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δύο πράγματα είναι σαφή. Καταρχάς, ότι σήμερα είναι λιγότερο δραστήριες οι οργανώσεις αυτές για την παρακολούθηση της κυβέρνησης και κατά δεύτερον, η πιο πολλή έρευνα περιορίζεται σε project που γίνεται σε τομείς από διεθνείς και όχι αλβανικές ε, ενώσεις. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ε, αυτές θέτουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς. Να αναφέρω κλείνοντας κάποιες βασικές συστάσεις για την Αλβανία. Χρειάζεται πολιτική θέληση και ομοφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων για να περάσουν οι αλλαγές. Να τεθεί και το θέμα της πολιτικής ασυλίας. Θα πρέπει οι εκλογές στην άνοιξη του 2011 να πληρούν τα διεθνή στάνταρ και τις συστάσεις του ΩΣΑ που έγιναν πριν από ένα έτος θα πρέπει να ξεκινήσει συνεργασία, θα πρέπει να ξεκινήσει μάλλον ε, πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση και του δικαστικού σώματο. Και νομίζω ότι κάπου θα τελειώσει ο χρόνο μου. Σα ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Ντερβίση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα. Ξεκινάει η συζήτηση. Εγώ δυστυχώ θα πρέπει να σα εγκαταλείψω θα ήθελα να παραμείνω. Άλλο συνάδελφο Κούκα θα προεδρεύσει και μετά θα συναγάγει τα συμπεράσματα. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Αντιπροσωπείας για τη Βοσνία, Ζεγοβίνη, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία. Από μένα ευχαριστώ και καλό σας βράδυ. Θα τα πούμε το πρωί. Αύριο μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα καλέσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα σας καλούσα εσάς, αλλά θα έλεγα να ρωτήσουν πρώτα οι βουλευτές τις ερωτήσεις, γιατί μπορεί να ρωτήσουν και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν πιο ορθολογικό να σας δώσω το λόγο στο τέλος, αφού υποβληθούν οι ερωτήσεις. Έχω αρκετούς ομιλητές στον κατάλογο. Βίκτορ Μποστινάρου είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω αυτή την εκδήλωση και θα ξεκινήσω Μπαίνοντα στο ψητό, θα μιλήσω απότομα για τη διαφθορά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά όχι μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι όταν μιλάμε για τη διεύρυνση, αυτό είναι ένα απόλυτο ευρωπαϊκό θέμα και θα είναι θέμα που θα ανησυχεί όχι μόνο τα, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις, κάθε χρόνο στις εκθέσεις ε, είναι αυτό το θέμα και στην αντιπροσωπεία. Στη διαφθορά τι σημαίνει. Διαφθαρμένοι άνθρωποι και εκείνοι που διαφθείρουν. Υπάρχει ο διαφθείρων και ο διαφθειρώμενος. Και συνήθως μιλάμε μόνο για τους διεφθαρμένους, λησμονώντας εκείνους που διαφθείρουν, που είναι εξίσου σημαντικοί και θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερον, είναι σημαντικό να διαρωτηθούμε τι πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντας υπόψη την διαδικασία διεύρυνσης και προσχώρησης και αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει για να αποφευθεί η διαφθορά και κυρίως να διακοπεί σχέση μεταξύ ε, εκείνων που είσαι σε ψηλό επίπεδο και με πολιτικές αποφάσεις με τη διαφθορά πρέπει να εξετάσουμε πρώτα από τι γίνεται. Πρώτα από όλα χρηματοδότηση των κομμάτων. Εδώ είναι η ρίζα πιθανότατα της ε, διαφθοράς σε, στο πολιτικό επίπεδο. Δεν βλέπω ακόμα καμία στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο θεσμικό διάλογο ε, που να αναφέρεται από το θέμα όσον αφορά τη συνεργασία στα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατείων, άλλο μεγάλο θέμα για τη διαφθορά, διότι συνήθω οι δωρεές οι χορηγίες και άλλα χρήματα που μπαίνουν στην προεκλογική εκστρατεία ε, χορηγούνται με κάποιους όρους που τίθενται. Πρέπει τελικά να συμμορφωθούν και να αποκριθούν στις υποσχέσεις που έδωσαν οι πολιτικοί όταν βρεθούν στην ε, κυβέρνηση. Και είναι εδώ μπροστά μας το θέμα, μετά η διαφάνεια. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δύο προαναφερθέντων τομέων, έχουμε μια στρατηγική Έχουμε απαιτήσει στο διάλογο που κάνουμε με τους εκπροσώπους των Δυτικών Βαλκανίων. Μέχρι τώρα, όχι. Μετά, τι γίνεται με τη συζήτηση και να τίθεται προαπαιτούμενο στη θεσμικό διάλογο το εξής. να καθοριστεί να καθοριστούν οι συγκρούσει συμφερόντων και να γίνει σωστό χειρισμό. Όχι απλώ μπλα μπλα και λόγια. Να τα σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να λησμονούνται. Και αποκάλυψη των ε, εισοδημάτων και των περιουσιών των δημοσίων ε, προσώπων. Όχι επίσημα, είναι κάτι που γίνεται και σε άλλα κράτη-μέλη. Και τα αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδενικά. Πόθεν έσχες λοιπόν. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν κατηγορούμε τους άλλους, ας δούμε εμείς τι κάνουμε πρώτα απ' όλα. Έχουμε πολιτικό διάλογο με διάφορα πολιτικά κόμματα της περιοχής. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει πριν η επαφή ή πριν μπει σε κάποιο μεγάλο κόμμα, μπει στο ΕΛΚ, στο Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα κλπ θα πρέπει το κόμμα αυτό να, τηρεί, να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών, βεβαίως, των προϋποθέσεων είναι τα κριτήρια για έλεγχο, για διαφάνεια, όσον αφορά την χρηματοδότηση του κόμματος, ε, προεκλογική εκστρατεία κλπ. Μέχρι τώρα, τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια στρατηγική ούτω ώστε να εφαρμοστεί αυτή συντονισμένα στην περιοχή. Μέχρι τώρα, τίποτα. Εμείς τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και εμείς οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο σχετικά με το τι θα πρέπει να προωθούμε στις συζητήσεις μας με τα πολιτικά κόμματα της περιοχής για να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαφάνειας, ελέγχου, τίποτα και τα, πώς σηματοδοτούν τα διάφορα ιδρύματα των πολιτικών, οι φορείς των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε κριτήρια. Τα κριτήρια μήπως πρέπει να εφαρμοστούν και στην περιοχή ως προαπαιτούμενο. Θες να έρθεις στην πολιτική μας οικογένεια Φερρυπίν. Θα κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Έτσι. Σ' αρέσει, δέχεσαι. Δεν σ' αρέσει, δεν δέχεσαι. Αυτοί αποφασίζουν, όχι εμείς. Θέλουν να έρθουν όμως αυτοί να έρθουν στην πολιτική μας οικογένεια και όχι εμείς να πάμε σε αυτούς. Λοιπόν, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε θεσμικό διάλογο σχετικά με τις πολιτικές μας σχέσεις με τους πολιτικούς φορείς της περιοχής. Εγώ να αναφέρω μια και μόνο περίπτωση. Την Αλβανία, την αλβανική υπόθεση. Εδώ και τις εβδομάδες ξέσπασε τεράστιο σκάνδαλο ε, διαφθορά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Κατηγορίες αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, η κυβέρνηση κατηγορούσε την υπολίτευση, καμία συνέπεια μέχρι σήμερα. Αλλά όσον αφορά αυτό το θέμα, οι δύο πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, η δική μου, το SND και το ε, ΕΛΚ, ακολουθούσαν, ταυτιζόταν, ε, μεροληπτούσαν κομματικά χωρίς να βλέπουμε ποιο είναι προς συμφέρον της Αλβανίας να προετοιμαστεί ούτως ώστε η Αλβανία τελικά να μπορέσει να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σίγουρα μπορούμε. Αλλά είναι σημαντικό όχι μόνο να κατηγορούμε τους εκπροσώπους των Δυτικών Βαλκανίων και να μην κοιτάμε τι γίνεται στην αυλή μας και να μην κάνουμε κάτι που είναι πανεύκολο να γίνει. Και στο τέλος και ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα πώς να το πούμε, στατική είναι υπερβολικό. Αλλά θα έπρεπε να συνεργαστούμε για να καταρτήσουμε κάποια κριτήρια που θα είναι προαπαιτούμενα για το διάλογο με τους πολιτικούς ηγέτες, κυβερνήσεις, κοινωνίες των πολιτών της περιοχής. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό θα εξακολουθούμε να συζητάμε για το ίδιο θέμα, όχι μόνο του χρόνου. Αλλά μέχρι σώτου τελειώσει η διαδικασία της διεύρυνσης. Και μετά θα συζητάμε ξανά μανά διαφθορά με τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς να λύνουμε τα προβλήματα και πολλά από τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μόλις 35 λεπτά μας έχουν απομείνει και 7 ομιλητέ ε, στον κατάλογο των αγορητών. Θέλω να ακούσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλω να ακούσουμε και τους τρεις επιφανείς προσκεκλημένους μας. Δεν θα σας θέσω όριο χρονικό, αλλά απευθύνω έκκληση στην υπευθυνότητά σας και στην αυρότητά σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στον κύριο Σαλαβράκο, που είναι και Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη Μακεδονία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και πρώτα απ' όλα θέλω να χαιρετήσω την ε, πρωτοβουλία της Προεδρίας της Επιτροπής και της Γραμματείας για το θέμα το οποίο έφερε σήμερα. Το οποίο δεν είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής βέβαια, αλλά είναι ένα θέμα μίζωνος κοινωνικού προβληματισμού, το οποίο θα μας βοηθήσει να παίρνουμε αποφάσεις για εξωτερική πολιτική. Απεκόμισα την εντύπωση ότι θα φύγω από αυτή την έδωσα όπως θα έφευγα από μια κηδεία. Ξέρετε, μετά τις κηδείες όλοι πιστεύουμε, βλέπουμε τη ματαιότητα των πραγμάτων και όλοι λέμε τι μάταια είναι η ζωή. Την επομένη όμως συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό τη ζωή μας. Εάν είναι να μείνει έτσι για όλους μας αυτή η συνάντηση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα θα έχει αν μας δημιουργήσει τέτοιο προβληματισμό ώστε αυτά τα οποία είπε ο φίλος μου ο κύριος Μποστινάρου να τα προχωρήσουμε, να τα μελετήσουμε και να τα επεκτείνουμε. Διότι, ως φαίνεται, η ανθρώπινη φύση ρέπει προς την παρανομία. Μια μικρή παρανομία έγινε και εδώ που ακούστηκε ότι υπάρχει εκπρόσωπος της Μακεδονίας, δεν υπάρχει Μακεδονία ανεγνωσμένη παρένθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι φύρο. Άρα ανεχόμεθα παντού τις παρανομίες, τις μικρές και τις μεγάλες. Η ανοχή αυτών των ε, παρανομιών από όλους μας δημιουργεί ένα χαλί πάνω στο οποίο περνάει και η διαφθορά. Μας είπαν οι κυρίες και ο κύριος από την Αλβανία, ο κύριος Δερβίσης, τα ίδια σχεδόν πράγματα. Τα ίδια σχεδόν πράγματα τα οποία λέει η Διεθνής Διαφάνεια, η οποία έβγαλε χθε το πόρισμά της. Και διαρωτώ με, τα Βαλκάνια είναι μόνο διεφθαρμένα κυρίε και κύριοι συνάδελφοι ή όλος ο κόσμος είναι διεφθαρμένος. Διότι εδώ από τη διεθνή διαφάνεια προκύπτει ότι όλη η ανθρωπότητα είναι διεφθαρμένη πλέον. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μια κόλαση του Δάντε. Πιο διεφθαρμένοι ποιοι είναι. Τα πολιτικά κόμματα, κατά τις απόψεις των πολιτών και των στατιστικών, οι δημόσιοι υπάλληλοι, η δικαιοσύνη, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την άσκηση εξουσίας ιδιαίτερα κρατικής. Υπάρχει όμως, στον... αυτό συμβαίνει στα λιγότερο προηγμένα κράτη. Στα περισσότερο προηγμένα κράτη, ποιοι είναι η διαφορά, είναι οι μεγάλες εταιρείε. Τι συνέβη με, ο... με ορισμένες μεγάλες εταιρείες ευρωπαϊκής προελεύσεως στην Αμερική, σε, άλλα, ε, σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, δεν υπήρξαν τάσεις και υποθάλψεις διαφθοράς, διότι όπως είπε και ο φίλος μου ο κύριος Μποστινάρου, διαφθαρμένος είναι αυτός που δίδει και αυτός που παίρνει. Λοιπόν, εάν συνεχίζουμε να υποκρινόμαθα δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα διότι το πρόβλημα αυτό θα μας οδηγήσει σε μίζονες ταλαιπωρίες μελλοντικά. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτές οι χώρες των Βαλκανίων είναι υπό εξέταση στο μικροσκόπιο και να μην βλέπουμε και να βλέπουμε εκεί μικροσκοπικά τα, τα μικρά μικρόβια και να μην βλέπουμε τα μεγάλα μικρόβια τα οποία είναι διαγυμνού οφθαλμού ορατά εις όλη την Ευρώπη. Παρακαλώ λοιπόν να επαναληφθεί αυτή η συνάντηση εις τρόπον ώστε να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη λύση του θέματος διαφθοράς ή για την βελτίωση των συνθήκων σε όλη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στα Βαλκάνια, υπό τις οποίες θα κάνουμε τη διαφθορά να μειωθεί. Διότι εάν μείνουμε έτσι δεν θα κάνουμε τίποτα. Με εκπλήσει όμως το γεγονός όσον αφορά τα Βαλκάνια ότι το περίεργο είναι ότι εκεί ενώ έχουμε εθνικιστικές εξάρσεις έχουμε παράλληλα και διαφθορά. Ξέρετε, οι εθνικές, εθνικιστικές εξάρσεις είναι κάτι το ιδεώδες. Λιμπερτέ, γκαλιτέ, φλατελιτέ και παράλληλα διαφθορά. Το είδαμε και στη Γαλλική Επανάσταση, το βλέπουμε και τώρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είμαστε τελικά και τι υποθάλπουμε τελικά. Θα σταθούμε στην τήρηση των νόμων ή θα κάνουμε μια ακαδημιακή συζήτηση τύπου λέσχης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Το λόγο έχει ο κύριος Ζόραν Τάλερ, ο εισηγητής για τη Μακεδονία, λέει ο πρόεδρος και πάλι. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου για τη διοργάνωση της σημερινής ακρόασης και να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας και να τους συγχαρώ θερμά για το θάρρος, για το κουράγιο που έδειξαν με την έλευσή τους εδώ. Δεν θα ήθελα να παρανοήσετε την ερώτησή μου. Θα ρωτούσα την κυρία Τσάλοβιτς, αισθάνεται απειλούμενη στη χώρα της, γιατί μας περιγράψατε ένα μαυροβούνιο, μια χώρα που δεν επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση, ιδιαίτερα την τολμηρή έκφραση όπως ε, η δική σας. Αισθάνεστε, αισθάνεστε να, να απειλείτε η ζωή σας στην πατρίδα σας. Στη διαφθορά υπάρχει η δωροδοκία και η δωροληψία είναι να δούνε και λαβή. Αυτό ισχύει όχι μόνο στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και σε πολλέ χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα νοοτροπία, είναι θέμα πελατοκρατίας, ευνοιοκρατία, ρουσφετολογία. Είναι νοοτροπία αυτή. Κάποιο σκέφτεται, εγώ έχω την εξουσία, είμαι αρχή, θα εκμεταλλευτώ και θα καταχραστώ τη θέση μου όσο μπορώ. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας της ηθήνουσας τάξης. Δεν έχει σημασία μόνο ότι κάποιος είναι στην εξουσία. Είναι στην εξουσία και αμέσως ενδιαφέρεται να εισπράξει. Μιλάμε για μια διαπλοκή των, ε, του οργανωμένου εγκλήματος, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ε, του δικαστικού κλάδου. Είναι ένα μόρφωμα ένα δίκτυο, ένα ολόκληρο κύκλωμα διαφθοράς και το στοιχείο κλειδί στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Θα πρέπει να φυπνίσουμε την κοινωνία των πολιτών για να αναλάβει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Κυρία Τάσεβα και κυρία Τσάλοβιτς, είστε ένα καταπληκτικό παράδειγμα εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με ένα κέριο θέμα, με ένα καθόδε ζήτημα στις ε, χώρες τους. Η πιο αδύναμη χώρα είναι η χώρα που περιλαμβάνει στην ε, εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω μία κέρια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι μέσα έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμήσει την ε, διαφθορά στις υποψήφιες χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που υψώνουν τη φωνή τους κατά της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για το Μαυροβούνιο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομο Γιατί και εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσάλοβιτς ε, κάποια θέματα. Γιατί ήταν ε, πολύ μεστή η παρουσίασή της ε, και ευρεία για τη φύση της διακυβέρνησης του Μοντενέγκρο στο Μαυροβούνιο και τα ίδια περίπου άκουσα και την περασμένη εβδομάδα από έναν εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης. Μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, αλλά και εκείνο ε, μου είχε εκφράσει αυτήν την διαγνώμη, διεφθαρμένοι, όλοι είναι ή μέλη της μαφίας ε, ή ανήκουν σε ένα κύκλωμα διαφθοράς, αλλά δυστυχώς ήταν μοναχική αυτή οι φωνή και απομονωμένη. Ούτε το διπλωματικό ε, σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε κάποιος πρέσβης επισήμαναν κάτι τέτοιο. Πώς εξηγείται αυτή η διαφορά σε ό,τι αφορά την αντίληψη για την κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Αναφέρθηκε επίσης το, τα ταξίδια που γίνονται πολύ συχνά και ποιος τα πληρώνει. Και είδαμε την ε, της έκθεση του Κοινοβουλίου και είδαμε ότι πολλά ε, ταξίδια τα πληρώνει το ίδιο το κοινοβούλιο. Μιλήσατε επίσης για την ιδιωτικοποίηση. Είπατε ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την ιδιωτικοποίηση ξοδεύτηκαν από την κυβέρνηση χωρίς να δώσει λογαριασμό. Έγινε η υπεξαίρεση αυτών των κονδυλίων από τα μέλη της κυβέρνησης και έχουν τοποθετηθεί σε ιδιωτικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Για παράδειγμα, πώς ε, εξόδεψε η ε, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου τα κονδύλια από την ιδιωτικοποίηση, αλλά αυτό είναι θέμα εσωτερικό. Θα πρέπει τα το κοινοβούλιο να αποφασίσουν αν χρησιμοποιήθηκαν σωστά τα κονδύλια αυτά, αν χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία υποδομών ή για να κλείσουν κάποιες ε, μαύρες τρύπες. Ναι. Αλλά όταν είπατε ότι τα χρήματα εκλάπησαν, υπεξαιρέθηκαν, υφαρπάχθηκαν ή δαπανήθηκαν ε, σε ακατάλληλου τομεί και όχι σε κατασκευή υποδομών, αυτό πραγματικά με σοκάρει. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ούλριχ Λούνατσεκ που είναι η συγκητρία για το Πέδιο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ εκτενείς και πραγματικά γλαφυρές εκθέσεις τους για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και την Αλβανία και Σιφοπέδη Μαυροβούνιο και την άποψη ιδιαίτερα της διεθνούς διαφάνειας. Όπως και προλαλήσαντες και εγώ μερικές φορές όταν ε, πηγαίνω στις χώρες αυτές και ακούω τις επικρίσεις για την εκτεταμένη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, έχω την αίσθηση όταν μιλώ ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλω να τους πω ότι και εμείς και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε λίγο ή πολύ διαφθορά και οργανωμένα έγκλημα. Σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αλλά η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα είναι φαινόμενο και στις ε, κοινοτικέ χώρες. Το θέμα είναι πώς θα διδαχθούμε από την εμπειρία μας. Το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων, της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατιών επίσης είναι θέμα. Μερικές χώρες έχουν ε, σημειώσει πρόοδο, εντυπωσιακή πρόοδο για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για το τι χρήματα δορίζονται ή τι χορηγίες δίνονται στο α ή β Αλλά στην πατρίδα μου δεν είναι όλα αυτά, δεν γίνονται όλα αυτά ξεκάθαρα και στο φως της δημοσιότητας. Εκεί λοιπόν πολλές χώρες θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε σε ό,τι αφορά αυτή τη διαφάνεια. Έχω κάποιες ερωτήσεις. σε Μία παρόμοια με αυτή του Ζόραν Τάλερ. Όταν η κυρία Βάνια Τσάλοβιτς ε, ανοιχτά επέκρινε την κυβέρνηση της πατρίδας της, προβληματίστηκα ε, πώς χειρίζεται το θέμα στη, στο Μαυροβούνιο. Αισθάνεστε φόβο, αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πατρίδα σας με αυτό το ανοιχτό τρόπο με τον οποίο μιλάτε. Επίσης, το έργο της μη σα οργάνωση ε, επικρίθηκε. Έγιναν ακροάσει στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, για παράδειγμα, όπου μπορείτε να επικρίνετε ανοιχτά την, ε, την κυβέρνηση. Επίση μιλήσετε για την έλλειψη κοινοβουλευτικού ελέγχου, την αδυναμία του Κοινοβουλίου να ελέγξει την κυβέρνηση. Όταν εσεί, μιλάτε έξω από τα δόντια και το ίδιο έκανε δεν βρίσκω το όνομά τη ή το όνομα του. Το ίδιο έκανε και ο κύριο ε, Λούτφι Ντερβίση. Γίνεται δημόσια συζήτηση ή ε, κοινοβουλευτική συζήτηση για τα θέματα αυτά στην Αλβανία. Υπάρχει ένας τρόπος για ανοιχτή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ώστε να αφυπνιστεί και η κοινωνία, το ευρύ κοινό, να ευαισθητοποιηθεί ο, ο κόσμος. Επίσης, ε, πώς, ε, τι απήχηση έχετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε καταρχήν φωνή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας σας. Έχετε κάποια προβολή. Έχετε δυνατότητα να εκφραστείτε εκεί. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι τα περισσότερα στοιχεία για την έκθεση πρόοδου της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα συγκεντρώνει από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την κατάσταση στη χώρα. Οπότε ελπίζω ότι και οι δικές σας εκθέσεις εξετάζονται με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Επιτόπου. Ισχύει αυτό? Έχετε κάποια δυνατότητα τροφοδότησης με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την εμπειρία σας. Το θέμα της κοινωνίας των πολιτών, ανάγκη ανεξαρ... ανεξαρτήτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ανεξάρτητες οργανώσεις που θα έχουν το κουράγιο, το χρόνο, την ενέργεια, την πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και τα χρήματα για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους, σαν αυτό που κάνετε εσείς και που είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και φυσικά χρειαζόμαστε και ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και αυτό το πρόβλημα έχουν πολλές χώρες. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να μου πείτε. Ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι μερικοί από εμά είμαστε εισηγητέ των εκθέσεων για τι πατρίδε σα. Εσεί τι περιμένετε από εμά, τι θέλετε από εμά όταν θα συναντηθούμε με εκπροσώπου τη κυβέρνηση κατά την εκπόνηση των εκθέσεών μα. Είστε καταρχήν ικανοποιημένοι από τι εκθέσει που συντάσσουμε. Είστε ικανοποιημένοι από τι δημόσιε δηλώσει μα ή από τι επισκέψει που πραγματοποιούμε στη χώρα σα. Θέλετε να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί, πιο επικριτικοί, να τα λέμε κι εμεί ε, πιο μάκια έξω από τα δόντια. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σας ευχαριστώ. Το λόγο του Θα είμαι σύντομο. Σε αυτή τη συζήτηση δεν θα ήθελα να ακολουθηθεί μια προσέγγιση που λέει πόσο είναι διεφθαρμένοι, κανένας δεν είναι διεφθαρμένος, όλοι είναι ένοχοι, κανένας δεν είναι ένοχος. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέτουμε στόχους και πάνω απ' όλα τα στάδια για να φτάσουμε σε μια μείωση της διαφθοράς. Εάν δούμε τη χθεσινή ταξινόμηση μπορούμε να συζητήσουμε πολλά όσον αφορά την Ευρώπη και αυτό το φαινόμενο συνοδεύεται νομίζω από κάτι απλούστατο παρόλο που τελικά είναι δύσκολη αντιμετώπιση, περίπλοκη. Έχουμε εκθετική αύξηση της διαφθοράς όταν υπάρχει επιδείνωση της εφαρμογής των κανόνων και βασικοί δημοκρατικοί πυλών σε μια χώρα διαβρώνονται. Όταν αυτό συμβαίνει γενικά ε, εξαπλώνεται και αυξάνεται η διαφθορά. Και υπάρχει μια μικρή διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και εκείνων που θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί κατά κάποιο τρόπο υπάρχει δυνατότητα μιας ανανέωσης ή αλλαγής της κυβερνήσεως. Σε κάποιες χώρες, στο Μαυροβούνιο, πόσα χρόνια ε, είναι που έχουν αυτή την κυβέρνηση. Είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ ήθελα όμως να κάνω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Κατά την άποψή σας η ευρωπαϊκή παρουσία και των διεθνών οργανώσεων άλλαξε, βελτίωσε ή όχι τα στοιχεία όσον αφορά τη διαφθορά. Ε, γιατί αυτό είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για να ξέρουμε αν η δική μας παρουσία εκεί χρησιμεύει ή δεν χρησιμεύει, αν βοηθάει για να βρεθεί απάντηση στα προβλήματα. Μιλήσατε για την αντίληψη που έχει ο πληθυσμό όσον αφορά την εκτεταμένη διαφθορά. Και γενικά όταν αυτό ε, επισημαίνεται είναι και μία ένδειξη καχυποψίας έναντι εκείνων που κυβερνούν σε διάφορα επίπεδα. Εγώ νομίζω ότι σαν κοινωνία των πολιτών κάνετε σημαντική ε, προσπάθεια, αλλά μερική κοινωνία των, τιματική ε, κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να ξέρουμε πόσο έχει δυσδύσει, έχει παρισφρήσει την κοινωνία των πολιτών διαφθορά, μέχρι ποιο βαθμό έχει δυσδύσει η διαφθορά. Διότι εάν έγινε ένα έθιμο, ε, ακόμα και η κοινωνία των πολιτών, παρά τις γενναίες προσπάθειές σας, ε, θα δέχεται αυτή τη δίσδυση. Είσαστε ένα μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Περιμένετε εσείς μια βελτίωση των συνθήκων με πλησίασμα στην Ευρώπη ή υπάρχει μια διαφορία στον κόσμο. Γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εξετάσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Τελευταίος είναι ο κύριος Κυρίλοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θα πρέπει να καλούμε ανθρώπους συχνά για να γίνεται ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων, ούτω ώστε οι περισσότεροι συνάδελφοι να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τις χώρες που συζητούμε αφορά και τις γειτονικές χώρες. Έχει σχέση και με το γεγονός ότι οι εγκληματίες προπολού έχουν διεισδύσει και εμείς στην Ευρώπη εξακολουθούμε να συζητάμε θέματα ολοκλήρωσης. Αυτοί έχουν ενωθεί από παλιά, είναι πιο αποτελεσματικοί. Και τι είναι ανησυχητικό, είναι πολύ δυνατή είναι ήδη πάρα πολύ ισχυροί. Πρέπει να σας πω ότι όλο το λαθρεμπόριο και η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικά, σημαντικές δίωδοι του λαθρεμπορίου και επιτρέπουν κάθε είδους διακίνηση. Και μετά πάει Σερβία, Μακεδονία, Λεομιλητής, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία, προς δυσμάς. Όταν λέω είναι ισχυρή, έγιναν πραγματικά ισχυρότατοι λόγω του εμπάργου που εφαρμόστηκε στη Ιουγκοσλαβία. Τότε δημιουργήθηκε μεγάλη ανατάραχη, αλλά και χωρίς το εμπάργο είναι αρκετά, θα ήταν αρκετά δυνατή. Ποιο είναι το σημαντικό. Ότι είναι κόμβοι κάποιες χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα, σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό. Θυμάμαι πριν μπει η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, επεκρίνεται και γιατί όχι. Αλλά θυμάμαι ένα Βρετανό συνάδελφο που είπε βάσει αυτών των κριτηρίων ένα κράτος μέλος που ήταν ιδρυτικό μέλος δεν θα μπορούσε να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι κοινή μάχη, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες σε χώρες που είναι κόμβοι. Δεν είναι πραγματικά μεγάλες χώρες Είμαι ευγνώμων για τις πληροφορίες που έδωσε η κυρία. Από παλιά ήξερα ότι το Μαυροβούνιο ήταν τέτοιος κόμβος και το ότι αυτή η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι ε, στην εξουσία επί μακρόν δεν είναι τυχαίο. Ας το δούμε, είναι αδύνατον κάτι τέτοιο. Η εξουσία αυτή, η ισχύς στην κυβέρνηση χορηγείται το οργανωμένο έγκλημα. Και αν δεν συγκεντρωθούμε και αν δεν δράσουμε δεόντως θα έχουμε πολλά βάσανα. Αναφέρθηκε το θέμα του κοσυφοπεδίου προηγουμένω. Βλέπουμε την αστάθεια ακόμα και τώρα στο κοσυφοπέδιο. Πολιτική αστάθεια σε ύψιστο επίπεδο. Γιατί? Μπορούμε απλώς να μαντέψουμε, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι το μεγάλο χέρι του οργανωμένου εγκλήματος. Η χείρα του εγκλήματος, των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που κάνουν ό,τι τους κατέβει στο, στο τι ό,τι θέλουν. Υπήρχε μια περίπτωση όπου τρεις Γερμανοί, τυχαία, κατηγορήθηκαν ως τρομοκράτες. Αυτοί τρεις Γερμανοί ερευνούσαν ένα έγκλημα διαφθορά σε στο επίπεδο. Τώρα, πώς ξαφνικά συνελήφθησαν στο Κωσυφοπαίδιο, φυλακίστηκαν και κατηγορήθηκαν ως τρομοκράτες ότι ήθελαν να την ενάξουν, ξέρω εγώ, κάποια αποστολή του ΟΗΕ. Δεν είναι τυχαία αυτά. Δημιουργείται αστάθεια τι τρόπο και θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα σε πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να είναι προσεκτική όταν προβαίνει σε αξιολογήσει και αποτιμήσεις που δεν είναι πραγματικέ, όπω είδαμε και με το Μαυροβούνιο. Και ίσω εμεί θα πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικότεροι όσον αφορά το ρόλο μα, διότι μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά εμεί και όποτε συζητούμε ζητούμε αντιπροσωπείες, επισκέψεις και όταν πηγαίνουμε σε αντιπροσωπείες και κάνουμε επισκέψεις πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί και ρεαλιστές. Αλλά λέμε ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Όπως μας την περιέγραψε η φιλοξενούμενη μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυρίλοφ. Και τώρα ο κύριος Μαραγκός, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Χαίρομαι ιδιαίτερο για τη σημερινή μου παρουσία εδώ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά γιατί βρίσκομαι μεταξύ φίλων και συναδέλφων που είναι όλοι αφοσιωμένοι στο στόχο της υλοποίησης σταθερών αποτελεσμάτων και από των αποτελεσμάτων στον πολύ σημαντικό αυτό τομέα. Θα ήθελα να πω ευθύ εξ αρχή ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πρωταρχική προτεραιότητα της ε, πολιτικής διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι καινούργια προτεραιότητα. Την καλύπτουμε το θέμα, την καλύπτουμε τη διαφθορά και στις εκθέσει προόδου και στο διάλογο με τις χώρες και με τα προγράμματα ΕΠΑ. Και έχω και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, μόνο το 2009 δώσαμε 80 εκατομμύρια σε, θέμα, σε προγράμματα κράτους δικαίου για την πάταξη της διαφθοράς, τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου. Είναι σημαντική πυλώνες η αστυνομία και η δικαιοσύνη για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και από το 2007 σε όλες τις χώρες ε, χρηματοδοτήσαμε προγράμματα αξίας 30 εκατομμυρίων μόνο και μόνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Και το πιο σημαντικό δεν είναι το ποσό, ο αριθμός. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συντονισμένη προσέγγιση και μια πολιτική βούληση και δέσμευση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο είναι η ανανεωμένη συνένεση για τη διεύρυνση του Δεκεμβρίου του 2006. Συμπεράσματα του Συμβουλίου ανέφεραν τη, με, τη μέρημνα των κρατών μελών από τα διδάγματα της πρόσφατης διεύρυνσης ότι το κράτος δικαίου θα πρέπει να είναι σημαντική προτεραιότητα σε προκαταρκτική φάση της ενταξιακής διαδικασίας. Οπότε χώρες που προσβλέπουν στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεσπίζοντας ένα πλαίσιο αλλά και εφαρμόζοντά το ήδη από τις πρώτες φάσεις της ενταξιακής διαδικασίας. Και αυτό είναι κάτι που παρακολουθούμε ετησίως με τις εκθέσεις πρόοδου και φέτος θα υποβάλουμε τις δύο γνωμοδοτήσεις μας για την Αλβανία και το Μαυροβούνιο για θέμα, και το θέμα της πάταξης διαφθοράς θα έχει κεντρική θέση. Είναι από τα σημαντικά πολιτικά κριτήρια και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το κεφάλαιο 23 ασχολούμαστε με τη μυθοδολογία, με αρχικούς και τελικούς συγκριτικούς κανόνες. Έχουμε πολλά ισχυρά εργαλεία και μηχανισμούς γι' αυτό. Καταρχήν την ενταξιακή διαδικασία που είναι ένα έναυσμα είναι ένα σημαντικό μέσο που ευνοεί και επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες. Ενδιαφέρει και τους πολίτες και αν λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες των πολιτών, σίγουρα οι πολίτες περιμένουν με το που θα ενταχθούν στην Ένωση να έχουν λιγότερη διαφθορά. Βέβαια κάποιοι θα υποφεληθούν από την δωροδοκία και τη διαφθορά, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό η πλειοψηφία των πολιτών πλειοψηφία τη κοινή γνώμη είναι κατά τη διαφθοράς. Οπότε είναι σημαντικό αυτό ο στόχο. Χρηματοδότηση των κομμάτων. Έγιναν πολύ εύστοχα σχόλια από τον κύριο Μποστινάρου. Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και πρότυπα εδώ. Μα ενδιαφέρουν οι βέλτιστε πρακτικέ. Και αν διαβάσετε προσεκτικά τι εκθέσει των τελευταίων χρόνων, έχω τι εκθέσει για την Αλβανία και το Μαυροβούνιο, και εκεί τα θέματα αυτά αναφέρονται κατά προτεραιότητα. Και μάλιστα όχι μόνο τυπικά, όχι μόνο στα λόγια. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η τυπική ύπαρξη των νομοθετικών διατάξεων. Η επίβλεψη, η επιτήρηση ήταν ελαττωματική στο Μαυροβούνι. Υπάρχουν εποπτικές αρχές, αλλά δεν ασκούν δεόντως επαρκώς την επιτήρηση. Μια το Υπουργείο Οικονομικών, μια κεντρική εκλογική επιτροπή, μας ενδιαφέρει ένα πάγιο σύστημα, ένα εύρωστο σύστημα που θα λειτουργεί με υψηλές ηθικές προδιαγραφές. Και αυτού του είδους ο διάλογος και η δέσμευση των πολιτικών δυνάμεων της Ευρώπης μπορούν να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουμε. Πάντως το σημαντικότερο ζήτημα είναι η ανάμειξη και των εμπλεκομένων αρχών στις ε, χώρες και το πλαίσιο υπάρχει στις περισσότερες χώρες. Θα θέμα να ενισχυθούν οι ανεξαρτητές αρχές, να, εξα... να ενισχυθούν οι εποπτικές αρχές, να κλείσουν τα παραθυράκια του νόμου, οι κερκόπορτες, γιατί πολλές φορές ε, η κατάρτιση των δικαστών μπορεί να μην είναι σωστή ή να μην εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Εμείς προσφέρουμε αρρωγή και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εκπροσωπούνται εδώ έχουν ε, λάβει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, για να αφυπνίσουν την κοινωνία, για να ασχοληθούν με συγκεκριμένους τομείς όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, ιδιωτικοποίηση, φορολογία κτλ, δικαστική, δικαστικός κλάδος. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα απτά αποτελέσματα και με την ανανεωμένη συνένεση του 2006 και με τη σεντόρια φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητά έμπρακτη μεταρρύθμιση και απτή μεταρρύθμιση και όχι μόνο τυπική μεταρρύθμιση ε, στα χαρτιά και στην νομοθεσία ε, με νομοθετικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε αποτελέσματα που θα έχουν διάρκεια. Έχουμε και σχετική ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και θα εκπονήσουμε στην Γενική Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων ένα πακέτο, μια δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα υποβάλλουμε το 2011, αλλά για τη διεύρυνση με τα πολιτικά κριτήρια και με την υποστήριξη όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα και να ενθαρρύνουμε τις χώρες να πραγματοποιήσουν ε, αισθητή πρόοδο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρίε και κύριοι. Ακούσαμε κάποια ενδιαφέροντα και σαφή σχόλια από τους αξιότιμους προσκεκλημένους. Ακούσαμε και τις σαφείς ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτέ. και τώρα θα ήθελα να ακούσω τις σαφείς απαντήσεις στα σαφή αυτά ερωτήματα. Να δώσω το λόγο τον κύριο Τερβίση. Μετά να ακούσουμε την κυρία Τσάλοβιτς και τέλο την κυρία Τάσεβα. Κύριε Τερβίση, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο Για το ερώτημα της δημόσιας συζητήση. Ναι, γίνεται δημόσια συζήτηση, αλλά όπως είπε ο κύριο Μαντσέρη, όλοι κατηγορούνται ε, για διαφθορά. Τελικά κανένα δεν είναι διαφθορμένο πολέμηση της διαφθοράς υποφέρει και πλήττεται από πολιτικοποίηση του θέματος στη χώρα μου από ασθενές δικαστικό σώμα. Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην τιμωρησία. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και έχουμε πολλά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν είναι ανεξάρτητα. Οι συντάκτες δεν μπορούν να λάμβανουν αποφάσεις βάσει επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά βάσει του τηλέφωνου που που δέχονται από τις ομάδες πίεσης. Χρειαζόμαστε πιο ασθενή πολιτικά κόμματα. Έχουν υπερβολική δύναμη στα χέρια τους τα πολιτικά κόμματα στην περιοχή μας. Πιο πολύ δύναμη από κάθε άλλο θεσμό στη χώρα. Και είμαστε βέβαιοι κατά κάποιο τρόπο ότι δεν κάνουν αυτά που κηρύττουν σε ό,τι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης, ε, για τις εξαρτήσεις τους και ούτε καθεξής και τέλος. Δεν χρειαζόμαστε έναν πόλεμο σε όλα τα μέτωπα κατά τη διαφθορά. Χρειαζόμαστε έξυπνες παρεμβάσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στον τομέα της υγείας. Χρειαζόμαστε επέμβαση στον τομέα της υγείας. Συγκεκριμένες δράσεις. Τέλος. να μην περιμένετε θαύματα σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο χρόνια. Γιατί αυτό είναι ένας από τους κινδύνους ε, της εργασίας ε, των ε, οργανώσεων κατά της διαφθοράς. Γιατί οι δωρητές περιμένουν αποτελέσματα σε έξι μήνες, ένα χρόνο. Αλλά είναι ένας πόλεμος που διαρκεί μια ολόκληρη ζωή. Και δεν μπορεί να κερδιθεί από μια κυβέρνηση, χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι οι φορείς.